σύνολο των μεγάλων καταστροφών ανά τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είδου συνέπειες θα έχει αυτή η απουσία ε, ρευστότητας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανθρωπιστική της δράση δεδομένων των φυσικών και άλλων καταστροφών που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι θα συμβούν το 2014. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα θα ήθελα καταρχήν, μιλώντας για τις προτεραιότητες για το 2013, να σας μιλήσω για το 12, διότι αυτό που συμβαίνει φέτος θα έχει άμεσες επιπτώσεις για το 2013. Το 2012 ασχοληθήκαμε με μία σειρά κρίσεων. Τρεις όμως είναι αυτές οι οποίες υπερβαίνουν σ' άλλες. Καταρχήν, η κρίση στο Σαχέλ λόγω της εξηρασίας και οι επιπτώσεις που υπήρχαν στη Λιβύη και στο Μαλί. Δηλαδή υπάρχει επίπτωση σε ολόκληρη την περιφέρεια αυτής της ευρύτατης ξηρασίας. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, ξηρασία έγκαιρα και μαζί με τον Επίτροπο Πίμπαλξ από τους πρώτους μήνες διαθέσαμε 337 εκατομμύρια ευρώ, επισύροντας την προσοχή στην κρίση στην περιοχή του Σαχέλ και ζητώντας ε, ε, ανθρωπιστική βοήθεια εγκαίρως. Δηλαδή εκεί όπου μπορούμε να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε την καταστροφή. Θυμάμαι έναν ανταποκριτή του BBC το Φεβρουάριο όταν ήμουν στο Τσάντ και στο Νίγηρα, που με ρώτησε «Κύριε Επίτροπε, πώς μπορείτε να μου ε, εξασφαλίσετε το ότι δεν θα βρίσκομαι εδώ σε έξι μήνες για να κινηματογραφώ παιδιά που ε, λιμοκτονούν». Και του απάντησα ότι θα ανταποκριθούμε σήμερα. Έτσι αποφύγαμε την κρίση, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε αποδυναμωμένους πληθυσμούς. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τρεις ξηρασίες σε 7 χρόνια και πολλές επιπλοκές που δημιουργούνται στο βορρά του Μαλή. Ήμουνα στη Μπουρκίνα δύο εβδομάδες πριν, ήρθα, ε, τον, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό τρεις μέρες πριν εκδιωχθεί. Και μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση στο βορρά του Μαλή επιδεινώνεται με τους εξτρεμιστές οι οποίοι πιέζουν ακόμα και τους Τουαρέγ έξω από μεγάλες πόλεις. Δεν μιλάμε λοιπόν για ε, στρατιωτικές μάχες, δηλαδή για το ότι μάχονται κατά του στρατού, ο οποίος είναι και ανύπαρκτος, αλλά Τη στιγμή που δεν είναι ενεργή η διεθνής κοινότητα, το, τα πράγματα επιδεινώνονται. Δηλαδή, το Μαλί, η κατάσταση του Μαλί θα ολιστήσει και στη Σομαλία. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις μπόρεσαν να δράσουν στο βορρά του Μαλί. Δηλαδή, δυσχερή η κατάσταση, αλλά αντιμετωπίσιμη μετά από πολλά χρόνια ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με την ευρύτερη κοινότητα. Αυτό θα είναι και προτεραιότητα για του χρόνου. Ως προς τη Συρία. Από το καλοκαίρι η Συρία έχει κινηθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τη στιγμή που βομβάρδισε ο Ασάντ το δικό του το λαό, τον ίδιο του το λαό, οι ανθρωπιστικές συνέπειες εντός Συρίας και για τις γείτονες χώρες είναι ολοένα και δυσκολότερες. Επέστρεψα χτες το βράδυ από μία επίσκεψη στην Ιορδανία και στο Λίβανο σε πολλές οικογένειες και είδα ότι εντατικοποιούνται οι μάχες στη Συρία και τη στιγμή που υπάρχει πολιτική ευθυγράμμιση της αντιπολίτευσης πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει στρατιωτική ευθυγράμμιση και ένα στρατιωτικό συνασπισμός. Είναι πολύ δύσκολο η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους ανθρώπους σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη καταστροφή από την κατάρρευση του οικονομικού ιστού της χώρας. Το ψωμί στοιχίζει 20 με 25 φορές περισσότερο από τα ε, καύσιμα και μέχρι και 40 φορές πάνω σε ορισμένες περιφέρειες. Έτσι, τη στιγμή που δεν υπάρχει προσβασιμότητα για τους υπεύθυνους της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουμε το Διεθνές προσωπικό που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Όχι επειδή δεν έχει θεωρήσει από τον Ασάντα, αλλά επειδή δεν μπορεί να εργαστεί. Και το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη καταστροφή και ανέχεια εντός και εκτός Συρίας. Και αυτό το είδα και στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Στην Ιορδανία χτες 1.300 άνθρωποι ε, πέρασαν τα σύνορα σε σχέση με τους 400 των προηγούμενων εβδομάδων. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι μέχρι τρεις μήνες πριν οι πρόσφυγες της Συρίας δεν συμμετείχαν στην σύραξη, τώρα δυστυχώς ε, εμπλέκονται, γιατί βομβαρδίζονται και οι καταβλισμοί τους. Για το Λίβανο και την Ιορδανία η κατάσταση είναι άκρος επικίνδυνη γιατί δεν υπάρχει κανένα είδος ε, εξισορρόπησης της κατάστασης από καμία πλευρά και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενεργά την κατάσταση. Τώρα θα πρέπει να προωθήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια και η άποψή μου από την Ιορδανία και το Λίβανο είναι ότι εντάξει δώσαμε 400 εκατομμύρια ευρώ, 120, και 120 από την ανθρωπιστική, ε, ένα μέρος από την Κομισιόν και το υπόλοιπο προήλθε από τα κράτη-μέλη. Όμως αυτά τα χρήματα δεν οδηγούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια διότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι δεν υπάρχει προβλεψιμότητα ως προς την προσέλευση των χρημάτων. Ε, έδωσα, σκιαγράφησα την κατάσταση στην κυρία Ζολή. Μία ε, οικογένεια ε, προσπαθεί να εξασφαλίσει την, την εγγραφή της και χρειάζεται έξι μήνες μέχρι να γίνει η, η καταγραφή των προσφύγων που περνάνε τα σύνορα. Δεν είμαστε έτοιμοι δηλαδή για αυτή τη μεγάλη ροή, την έκρηξη ροής των προσφύγων εάν ανακύψει. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, κάτι το οποίο μας οδηγεί σε θέματα ε, προϋπολογισμού. When I visited that it was taking a bad turn after the elections, uh, the country was now with M23 being uh, uh, in... Η κατάσταση στη δημοκρατία του Κονγκό έχει επιδεινωθεί εκτός και εντός Γκόμα. Υπάρχουν μεγάλες ε, μεταναστευτικές ροές. Στη δημοκρατία του Κονγκό προσπαθήσαμε να αναχαιτήσουμε αυτό το κλίμα επιδίνωσης ε, προσθέτοντας και ε, χρήση ελικοπτέρων για την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και πρέπει πολλές φορές να μπορούμε έγκαιρα να εκενώσουμε και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αυτή η εκένωση έγινε ε, πολλές φορές με τον δόκτωρα Μοκουέγγε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο όπου εργαζόταν. Ε, χρειάστηκε λοιπόν να απομακρυνθεί με ειδικά δικά μας ελικόπτερα. Δηλαδή προβλέπουμε κρίση επιδίνωση της κατάστασης το 2013 και δείχνει, όλα αυτά δείχνουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Έχει σημασία η έγκαιρη αντιμετώπιση της κρίσης και αυτό με οδηγεί στις προτεραιότητές μας για το 2013. Από πλευράς ε, επιχειρησιακής καθαρά, ως προς τις προτεραιότητες για το 2013 θα πρέπει εκεί που μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας να το κάνουμε. Μιλάμε για πολλές χώρες, ε, Συρία, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Σαχέλ, Κέρας της Αφρικής, Σομαλία και Πακιστάν. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Και η δημοκρατία του Κονγκό για τους λόγους που προείπα. Θα πρέπει να τονίσω ότι το 15 το 10-15% αφορά τις ξεχασμένες ε, κρίσεις, ας το πω έτσι. Δηλαδή, είμαστε ο βασικότερος δωρητής για κρίσεις οι οποίες δεν ε, φτάνουν στη, στον τύπο, όπως η, η, στο Σαχαράουι, για τους Σαχαράουι ή για την Κολομβία. Από πλευράς νομοθετικής ή πολιτικών προτεραιοτήτων καθαρά, Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που τονίσατε κι εσείς και μας ε, βοηθήσατε ιδιαίτερα. Τη νέα δηλαδή επισητιστική, ε, το σύμφωνο επισητιστικής ασφάλειας. Εμείς είμαστε ιδρυτικό μέλος αυτής της ε, σύμβασης η οποία θα τεθεί σε ισχύ, σε ισχύ άμεσα. Τον Ιανουάριο δηλαδή του 2013. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να καταδείξουμε ότι δεν τα έχουμε καταφέρει ως προς την αντιμετώπιση της ε, πείνας και της λιμοκτονίας. Μαζί με τον Επίτροπο Πίμπαλξ μιλήσαμε για ανάγκες και μια ανακοίνωση για θέματα διατροφής. Έχει σημασία το πώς θα ορίσουμε τις ε, προτεραιότητες και πώς θα τις μεταφέρουμε από έτος σε έτος. Ως προς τα βασικά στοιχεία εργασίας για το 2013, την προηγούμενη φορά που ήμουνα ενώπιον σας μιλήσαμε για τον κανονισμό ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Και σας είπα ειλικρινά ότι δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί ο κανονισμός άμεσα. Πρέπει να ενισχυθεί όμως και να γίνει πιο αποτελεσματικός. Και αυτό προβλήθηκε από τη διαδικασία διαβούλευσης. Θέλουμε λοιπόν να εξεύρουμε τρόπους για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε έναν κόσμο όπου αυξάνονται οι ανάγκες και δυστυχώς δεν υπάρχει, η, δεν υπάρχει επαρκής ικανότητα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το δίκαιο περί ανθρωπιστικής βοήθειας τη στιγμή που ο κόσμος παλινοδεί από ασύμετρες σειράξεις και για να το κάνουμε αυτό έχουμε προωθήσει μία επιγραμμική διαβούλευση, δηλαδή η, ανθρωπιστική, η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια, πώς θα κινηθεί προς το στόχο της. Μέχρι το Μάρτιο του 2015 προβλέπεται η διαβούλευση και στη συνέχεια θα συνταχθεί μία ανακοίνωση η οποία θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως προς την ανθρωπιστική μας δράση. Επίσης, ένα σχετιζόμενο θέμα είναι η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στα πλαίσια του προγράμματος δράσης. Όλες οι μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε επιβεβαιώνουν τη διαδικασία συνένεσης που είναι απολύτως αναγκαία. Ιδιαίτερα για να είμαστε ουδέτεροι και αμερόληπτοι στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα για, από πλευράς ε, Βόρειου ε, Μαλή και αυτό αφορά παράλληλα και την κατάσταση της Συρίας. Ελπίζω να μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε στο εγγύς μέλλον. Επίσης προβλέπεται το πρόγραμμα δράσης το οποίο λύγει το δεύτερο εξάμεινο του 2013 και προβλέπει ένα πρόγραμμα δράσης που θα συνεχίσει αυτή την ε, συνενετική διαδικασία. Θα ήθελα, ήθελα να αναφερθώ και στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια στα πλαίσια του εθελοντισμού και χαίρομαι διότι εσείς έχετε συνεισφέρει σε αυτό το 13 το 12 με συγχωρείτε, προωθήσαμε αυτή τη δράση και το 13 θέλουμε να πάρει σάρκα και οστά, έτσι ώστε το σχετικό άρθρο της Συνθήκης της Λισαβόνας να υλοποιηθεί, να πραγματοθεί, να μπορέσουμε δηλαδή να προβάλλουμε και προβλέψιμες εξελίξεις. Μας ενδιαφέρει δηλαδή και η κατάρτιση εθελοντών. Και φυσικά η νομοθεσία θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή μόνο αν υπάρχει κατάλληλη δημοσιονομική υποστήριξη. Όσον αφορά τη νομοθεσία για την προστασία των πληθυσμών, θα ήθελα να πω ότι το 2013 ε, θα είναι κρίσιμη χρονιά. Υπάρχει η εξωτερική αυτή διάσταση, διότι η δυνατότητα προστασίας των πληθυσμών έχει μεγάλη σημασία σε μεγάλες κρίσεις όπως ε, τις μεγάλες καταστροφές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δύο τρίτα πέρυσι αντιμετώπισαν ε, φυσικές καταστροφές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και η Επιτροπή σας έχει συνδράμει και θα εξακολουθήσει να συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση. Ως προς το ε, έργο συνέχειας και ανθεκτικότητας, το έχουμε δει και με τον Επίτροπο Πίμπαλξ, θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στο κέρας της Αφρικής, στο Ουαγκαντούγκου, δύο εβδομάδες πριν. Προβάλαμε ένα πρόγραμμα ε, αντιμετώπισης των αναγκών του πληθυσμού και στο Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής, αλλά το 13 θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει ε, δυνατότητα αντιμετώπισης έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένη ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Ως προς τη συνεκτική μας προσέγγιση, Υπάρχει ένα κοινό ανακοινοθέν μεταξύ Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου μέσα στα πλαίσια της συνεκτικής αυτής προσέγγισης για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και καταστροφές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε και θέλουμε να επιλύσουμε κρίσεις και να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης εκεί που γίνεται. Και αυτό αφορά και το ανθρωπιστικό σκέλος. Γι' αυτό συμμετέχουμε σε προγράμματα δράσης, αλλά επειδή θα πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι και ουδέτεροι, στα πλαίσια της, ε, των ανθρωπιστικών οργανώσεων, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο έργο αυτής της ανεξάρτητης ε, εργασίας και έχει ε, σημασία να δούμε και να εντοπίσουμε τους πυρήνες όπου υπάρχουν επίμαχα ζητήματα. Ως προς τα δημοσιονομικά μας, μέσα στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου προσπαθούμε να επισύρουμε την προσοχή σε δύο ζητήματα και σας τα αναφέρω και εδώ. Ως προς τον, ε, την πρόταση προϋπολογισμού είμαστε ιδιαίτερα συνετοί ως προς τις προτάσεις μας. Ζητήσαμε πολύ μικρή αύξηση στη βασική γραμμή ανθρωπιστικής βοήθειας της τάξης του 8,9%. Αυτό αφορά το 24% αύξηση που προτινόταν στο κεφάλαιο 4. Ζητήσαμε όμως ε, περισσότερα χρήματα στο αποθεματικό επίγουσας ανάγκης, διότι αντιμετωπίσαμε χρονιές όπου δεν χρειάστηκε αυτό το αποθεματικό επίγουσας ανάγκης. Είχαμε ορισμένες καλές χρονιές πολύ παλιότερα, όχι από, υπό την αιγίδα μου. Γι' αυτό θέλουμε μία αύξηση της τάξης του 8,9% και έχω ένα απλό μήνυμα να αποστείλω. Αν γίνουν περικοπές, κάτι το οποίο απέφχομαι, γιατί δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τη θέση μας στον κόσμο. Νομίζω ότι ένα 8,9% ε, δεν είναι και τίποτα είναι θέμα απλής οικονομικής λογικής. Αλλά μεγάλη σημασία για την ΤΕΒΕ και το Κοινοβούλιο είναι να προστατεύσετε το αποθεματικό επίγουσας ανάγκης. Προτείναμε 350 εκατομμύρια τα οποία περιορίστηκαν σε 280 δεν έχει και μεγάλη σημασία για τον προϋπολογισμό, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους που προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε κατάσταση επίγουσας ανάγκης. Μιλάμε για ένα 0,62% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμεληταίο το ποσό. Αλλά βοηθάμε 150 εκατομμύρια ανθρώπους όταν το χρειάζονται, αυτό το 0,62% και είναι και ό,τι πιο σημαντικό επιτελεί η Ευρώπη. Ελπίζω να μας υποστηρίξετε. Εμείς ζητάμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς το ελάχιστο και ζητούμε ευελιξία εκεί όπου πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Και ελπίζω να μας βοηθήσετε να προστατεύσουμε τους πληθυσμούς αυτούς. Ευχαριστώ. Η κυρία Στίφλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για μια πληρεστάτη παρουσίαση. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στην Επιτροπή μας. Συναντηθήκαμε και στο Στρασβούργο και είχαμε και εκεί επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων. Καταρχάς θα συμφωνήσω σε κάποιες από τις παρατηρήσεις σας η έκθεση Γκαρντίνη για την πρόταση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έγινε δεκτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η δική μας Επιτροπή συνδέεται με τη διαδικασία και ελπίζω ότι αυτές οι δύο, λυπάμαι που αυτές οι δύο τροπολογίες ε, οι δικές μου απορρίφθηκαν από την Αρμόδια Επιτροπή για την οικονομική βοήθεια στον τομέα της πρόληψης και της προετοιμασίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, ήταν η μία τροπολογία, και για τον προϋπολογισμό είχα πει το 50% του τίτλου 3 σχετικά με την ασφάλεια και διασφάλιση του δημοσιονομικού πλαισίου και 50% που να προέρχεται από το 4 η Επιτροπή αποφάσισε να το κάνει 70% και 30% αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία των παρεμβάσεων σε επίπεδο πολιτικής προστασίας γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στις υποανάπτυξη χώρες τα ποσά για την περίοδο 14 με 20 θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την πραγματικότητα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι θα καταθέσω εκ νέου τις τροπολογίες αυτές στην Ολομέλεια και ζητώ την υποστήριξη όλων. Τώρα για τον κανονισμό, ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να επιμείνουμε ότι ε, θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι παρεμβάσεις σε ε, πραγματικές οικονομικές ανάγκες και να ενισχύουν τις τοπικές ικανότητες και δυνατότητες. Πάντα σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο ένα και πιο δύσκολο και λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών είναι σαφές αυτός ο εθελοντικός κώδικας να συμπληρώνει τα μέσα τα οποία είναι ήδη υπάρχοντα. Ε, κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου λοιπόν το 2013 τα θέματα αυτά θα τεθούν. Το 2012 κυρία Επίτροπε ήταν μια χρονιά ευαισθητοποίησης για τον κατεπήγοντα χαρακτήρα και τη σύνδεση της ανάπτυξης με την, απασχόληση γενικότερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε επίσης και με το λεγόμενο το θέμα το επιμέρους του σώματος των εθελοντών είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εσείς οι ίδιοι πήγατε στο Ουαγκαντούγκου πρόσφατα, αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 12 η τοπική ε, προχωρά σωστά, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Τώρα για την ανθρωπιστική βοήθεια στα πλαίσια της δημοσιονομικής βοήθειας για το 14 με 20 για τον προϋπολογισμό του 2013. Υπάρχει μία μείωση των πιστώσεων πληρωμών για την κατεπίγουσα βοήθεια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, το οποίο μου φαίνεται ότι παρουσιάζεται πλέον με πολύ δύσκολους όρους. για τον προϋπολογισμό του 13 επαναλαμβάνει η κυρία Στίφλερ και για την πιθανή μείωση του προϋπολογισμού. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε, πώς βλέπετε τα πράγματα με λίγα λόγια. Με μεγάλη ευχαρίστηση ε, σας συναντάμε εδώ, σας φροντίζουμε κι εμείς ε, και νομίζω ήδη απαντήσατε στις ερωτήσεις τις οποίες θα θέλαμε να σας θέσουμε, αλλά κάποιες από αυτές θα τις θέσω εκ νέου. Είναι σαφές ότι σε ορισμένε χώρες βιώνουμε πολύ δύσκολες κατάστασεις που επηρεάζουν άμεσα την ανθρωπιστική βοήθεια και αφορούν την ζωή, θα έλεγα, χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο κάνουμε και για τα οράματα τα οποία έχουμε ε, και σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει ε, στο Πακιστάν, στα σύνορα ε, Ερυθρέας, Αιθιοπίας. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένες πολύ επικίνδυνες περιοχές του κόσμου είναι η μοναδική παρούσα. Συνειδητοποιούμε, εν πάση περιπτώσει, την παρουσία μας αυτή και την, τον θετικό της χαρακτήρα. Ε, για πρώτη φορά πήγε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Επιτροπή Τροφιμικής Βοήθειας της, ε, της Διεθνούς Οργάνωσης ε, στη Ρώμη. Είμαστε επίσης σε στενές σχέσεις με την Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και είμαστε προφανώς η μεγαλύτερη δύναμη στον τομέα των προγραμμάτων τροφίμων και ο ΦΑΟ ταυτόχρονα προσπαθεί να συνεργαστεί μαζί μας γιατί εργάζεται και αυτός προς τις ίδιες κατευθύνσεις με διαφορετικό τρόπο από μας. Θέλετε να μας μιλήσετε για τις σχέσεις με αυτή την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Πού βρίσκονται οι σχέσεις αυτές και τι ρόλο μπορεί να παίξει η ανθρωπιστική βοήθεια πλέον στην κατάσταση την οποία βιώνουμε. Τελειώνοντας, αν μου το επιτρέπει η Προεδρία, μία επιπλέον φράση. Εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ε, βοήθεια η ανθρωπιστική σε οικονομικά επίπεδα. Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η βοήθεια αυτή για τα χιλιάδες οικογενειών στον κόσμο. Υπάρχει κρίση, δεν πρέπει να την χειροτερεύσουμε. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Επίτροπε. Μας κάνατε μια εντυπωσιακή παρουσίαση θα έλεγα των προγραμμάτων σας και των διαπιστώσεών σας. Είμαστε ευτυχείς σαν Επιτροπή που σας έχουμε σαν Επίτροπο γιατί οι πεπιθήσεις σας, η ευκρίνεια έκφρασης και η αποφασιστικότητά σας έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το συγκεκριμένο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μια ευχή λοιπόν και ένα κοπλιμέντο ε, για ε, τα Χριστούγεννα. Τώρα δύο ερωτήσεις ε, ή μάλλον μια ευχή καταρχάς. Ελπίζω η προσπάθειά σας να μην αντιμετωπίζει εμπόδια, αλλά αντίθετα να βελτιώνεται από την ολοένα βελτιούμενη συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ελπίζω ότι σε έφετο χρόνο η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα καταλήξει στον ποιος είναι ο ρόλος της ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και θα καταστεί δυνατό επιτέλους να βρεθούν τρόποι σωστής συνεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μία ομάδα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη ε, εργάζονται σαν μία γραφιά, είναι όλοι ενωμένοι, ενώ εμείς δεν το κάνουμε ακριβώς έτσι. Ας πούμε η συνεργασία ανάμεσα στην ΤΕΦΚΟ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν είναι αυτή την οποία θα θέλαμε και γι' αυτό θα θέλαμε και η δική σας υπηρεσία να υποφεληθεί από αυτό. Και μία ερώτηση τώρα τελικά θα μπορούσατε να ήσασταν παρακαλώ λίγο πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τις ανησυχίες και δυνατότητες τις οποίες έχετε σχετικά με το Βόρειο Μαλί. Ε, δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω γιατί έχω μια άλλη συνεδρίαση, αλλά ο συνεργάτης μου θα καταγράψει αυτό που θα πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φιές, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τα καλά λόγια και τους επένους προς την Επίτροπο να τη συγχαρώ για αυτά τα οποία κάνει. Θα ήθελα να θέσω εκ νέου το θέμα του Μαλή. Νομίζω ότι αυτό το οποίο διεξάγεται εκεί είναι το, χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Καντάφη και την επιστροφή των ενόπλων του Αρέγ στην χώρα και με τον συνάδελφο Φρανσουά Αλφόνση συναντηθήκαμε τρεις φορές με τους εκπροσώπους του MNLA που είναι η ομάδα των Τουαρέγγι η οποία είναι περισσότερον μετριοπαθής και διαπιστώνουμε ότι είναι διατεθειμένοι να καταλήξουν σε μία κάποια συμφωνία με την κυβέρνηση του Νότου της χώρας εφόσον η κυβέρνηση αυτή σεβαστεί ε, την αυτονομία των Σαουάτ είναι κάτι το προτιμότερο να συμβεί κάτι τέτοιο από έναν τέτοιο πόλεμο, αλλά δυστυχώς οι σάλπιγγες του πολέμου έχουν αρχίσει να ηχούν με τις ανθρωπιστικές καταστροφές το οποίο, αυτό το οποίο θα επιφέρει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να θέσω εκ νέου και ένα άλλο θέμα, το της Δυτικής Σαχάρας, της Παλαιάς Ισπανικής Σαχάρας. Είναι μια χένουσα θα έλεγα κατάσταση η κυβέρνηση της Ισπανίας και όχι μόνο συνεχίζουν να βοηθούν τους πληθυσμούς στην Δυτική Σαχάρα. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι κάτι το οποίο δεν βελτιώνεται με τον χρόνο λόγω και της ευρύτερης πραγματικότητας στο Σαχέλ δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα θα μπορούσατε να μας πείτε πώς πηγαίνουν τα πράγματα και αν πράγματι υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της ε, κοινοτικής βοήθειας με διαφορετικούς τρόπους. Ε, κυρία ε, Γεωργίευα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ξεκινήσω με το θέμα του Μαλή, Ναι, και ο κύριος Μπέρμα πρέπει να φύγει. Μπίερμα πρέπει να φύγει. Οι συνθήκες από ανθρωπιστική έποψε στο Μαλί είναι πολύ σκληρές. Ε, μετά τη Σομαλία είναι η δεύτερη χώρα το Μαλί σε θνησιμότητα παιδιών στην ηλικία κάτω των 5. Δεύτερη μετά, το Μαλί, μετά τη Σομαλία. Και η κρίση στο βορρά έχει προξενήσει 400.000 εσωτερικούς εκτοπιστέντες 200 μέσα στη χώρα και 200.000 200 εντός της και 200.000 εκτό των σύνορων. Μπορεί να μην επισκέφθηκα με το Βόρειο Μαλί, αλλά επισκέφθηκα, μίλησα με πρόσφυγε στη Βόρεια Μπουρκίνα, κοντά στον Τόρι. σε ένα στρατόπεδο προσφύγων και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά αναλαμβάνουν την ε, εξουσία οι εξτρεμιστές. Ο νόμος της Σαρία επιβάλλεται κατά τον πιο φρικαλαίο τρόπο. τρόπο. Ε, μας είπαν ιστορίες ότι αν ε, πιάσουν κάποιον να καπνίζει, τον αποκεφαλίζουν, τον, ε, του, βράζουν το κεφάλι και μετά το ξανακολλάνε πάνω στο, στο πτώμα και βάζουν όλο το χωριό να παρακολουθεί αυτές τις σκηνές. Γι' αυτό όλοι φεύγουν τρέχοντας. Και αυτό που μας ανησυχεί επίσης είναι ε, ότι η κυβέρνηση του Μαλή βρίσκεται σε πλήρη απόγνωση Χρειάζεται υποστήριξη τώρα, διεθνή στήριξη τώρα. Ε, εγώ πήγα ένα Σάββατο εκεί, συνάντησα τον πρόεδρο, αναπληρωτή πρόεδρο καλύτερα και τον ε, εκτελώντα χρέη πρωθυπουργού και τον Υπουργό Ανθρωπιστικών αρμόδια για ανθρωπιστικά ζητήματα. Επικοινωνία μεταξύ του, του ασκούντος τα καθήκοντα Προέδρου και του ασκούντος τα, τα καθήκοντα Πρωθυπουργού δεν υπήρχε. Μεταξύ τους ε, ο Πρωθυπουργό μιλούσε μόνο για κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος για εθνοσυνέλευση ε, και για να σας δώσω μια ιδέα του πώς έχει διαμορφωθεί, πόσο κακό είναι δηλαδή το πολιτικό περιβάλλον. Ο Πρωθυπουργό ζητούσε τη βοήθειά μου. Και τι προτεραιότητα έχει, ξέρετε. Τι θα περιμένετε να ζητήσει ένας πρωθυπουργό μιας χώρας όπου το μισό, η μισή επικράτεια βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση και είναι η δεύτερη σε υποσυτισμό μικρών παιδιών μετά τη Σομαλία, ανά τον κόσμο. Τι μου ζήτησε. Συστήματα αφής για την ε, για τις ψηφοφορίες της Βουλής του Μαλή. Αυτό ζήτησε. Οθόνες αφής. Και η απάντησή μου ήταν, ε, α παίξω λίγο το συνηγορό του, διαβόλου, του διαβόλου. Μήπω θα ήταν κάπω πρόημο να είστε τέτοιο πράγμα. Την ώρα που έγινε το πραξικόπημα, λατήθηκαν όλα τα κτίρια, τα κυβερνητικά, αφαιρέθηκαν οι υπολογιστέ, δεν υπάρχουν καν αρχεία του κράτους αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια, μια βαθύτατη πολιτική κρίση πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος βέβαια μου άφησε μια καλή εντύπωση και έρχεται και στις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Ε, προσπαθούν να βρουν ένα δρόμο λοιπόν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Ο στρατός, ο στρατός του Μαλή. Έχει ένα, μια μερίδα πάρα πολύ ισχυρή που μόνο προβλήματα προξενεί και οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ αδύναμοι. Είδαμε πώς κάθονται οι φρουροί της προεδρικής φρουράς πάνω στο να κούρκουδα και τα χαφυλάνε τον πρόεδρο. Πολύ σοβαρές ανησυχίες λοιπόν έχουμε για το Μαλί. Για τις MNLA, για τις ομάδες των ατάκτων, ναι, είναι διατεθειμένοι να ε, διαπροβούν σε διαπραγματεύσεις. Και γιατί, γιατί τώρα τους πιέζουν από την άλλη πλευρά οι εξτρεμιστές και θα πρέπει ταχύτερα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, αλλά πάντως οι πάντες πιστεύω θα συμφωνήσουν πως θα χρειαστεί η στρατιωτική επέμβαση, η επέμβαση του στρατού ε, για να καταπολεμηθούν αυτοί οι οποίοι δεν δέχονται να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσει. Ο Ακή και ο Αμπού Χαράμ, ε, παραδείγματι. Ο Αμπού Χαράμ ιδιαίτερο δεν, δεν, δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση στρατική επέμβαση τι σημαίνει. Σημαίνει ενίσχυση του στρατού του Μαλή, ανάπτυξη του δυναμικού, ταχύτατα. Και ξέρουμε ότι όπως και να έχει, ανθρωπιστική κρίση θα προκύψει. Όπου υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις, υποφέρουν οι άμαχοι. Το ίδιο με την Μπουρκίνα Φάσο μιλήσαμε με τους υποευθύνου εκεί, μας είπανε ένα μαλλί θέλουμε, δεν θέλουμε δύο, δεν θέλουμε να διχοτομηθεί. Βεβαίως έστω στο βορρά να έχουν πιο πολύ ανεξαρτησία και αυτονομία και πιο πολύ φεβασμό, αλλά μία να είναι χώρα και ενιαία. Αν μου επιτρέπετε τώρα θα περάσω στην κυρία Στρίφλερ, να ξαναρχίσω από την αρχή της ερωτήσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Καταρχάς, ο συσχετισμός της ανακούφισης της πρώτης ανάγκης, δηλαδή, με την ανοικοδόμηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και άλλωστε έχει να κάνει και με τις δικές μας προσπάθειες για την ανθεκτικότητα των κοινωνιών. Έχω πέραν του Αζίρ και του Σέρ εντοπίσει άλλες δύο ε, χώρες, την IT, καταρχάς, την οποία θα επισκεφθώ τον Ιανουάριο, στις 12 του μηνός για την τρίτη ε, επέτειο του σεισμού μέσα σε μια γενικότερη προσπάθεια της διεθνούς οργάνωσης μετανάστευσης για να αποδείξουμε ότι όλοι εκείνοι που ζουν σε στρατόπεδα ε, σεισμοπαθών τώρα μπορούν να, ε, να μετεγκαθίστανται σιγά σιγά σε πιο, μόνιμες, σε πιο μόνιμα καταλήματα και ο πρόεδρος Μπάσερ έχει δείξει πάρα πολύ καλό έργο, έχει δώσει 50 εκατομμύρια για τη στέγη, έχει επιτρέψει αυτό το συσχετισμό. Το ίδιο βέβαια και στην ακτή του Ελεφαντοστού, τη λεγόμενη Côte d'Ivoire. Έχουμε καλή πρόοδο μαζί με τον Επίτροπο Πίμπαλξ για την μετάβαση, όπως τη λέμε, για την εταιρική σχέση και τη μετάβαση μαζί με την ε, κυβέρνηση και την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, Γενική Διεθνή Ανάπτυξη. Αλλά καλά το επισημαίνετε, κυρία Στρίφλερ, το Αζίρ, το Σαχίλ, όπου ουσιαστικά δοκιμάζεται η ικανότητά μας να συσχετίσουμε, να συνδέσουμε την ανακούφιση με την ανάπτυξη. Την άμεση επέμβαση δηλαδή με την ανάπτυξη. Έχουμε ένα καλό πρόγραμμα ε, από τη βάση προς τα άνω, στην Μπουρκίνα Φάσο, τον Ήγυρα, το Μαλί βέβαια, αν και εκεί πολλά πράγματα όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να γίνουν. Έχουμε όμως ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, διότι πρέπει πάνω απ' όλα να αλλάξει η νοοτροπία και σε επίπεδο ανθρωπιστικής και σε επίπεδο αναπτυξιακής πολιτικής για την Μπουρκίνα Φάσο και την ε, ανακούφιση, πρέπει να σας πω, σε μια επίσκεψή μου είδα ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί ε, βρήκαμε ένα πολύ καλό τρόπο να καταπολεμήσουμε και τον υποσυτισμό με βραδίας μορφής επιδοτήσεις που επιτρέπουν ε, την εξασφάλιση επαρκούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα παιδιά με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Δηλαδή, την ώρα που, ε, την ώρα έπρεπε να πληρωθεί κάποιο, κάποια αμοιβή ιατρική, έχει καταργηθεί για τα παιδιά κάτω των 5 με πολύ ψηλή θνησιμότητα στην Πουρκίνα. Τη στιγμή όμως που μπορεί να πάει ένα παιδί στο γιατρό εγκαίρος, κερδίζουμε πολλά, εξοικονομούμε πολλά από την ανάγκη, από τα έξοδα για την θεραπεία εκ των υστέρων. Φόσο προληπτικά μπορούμε να δράσουμε, κερδίζουμε πολλά, πολύ περισσότερα από την θεραπεία. Αυτά λοιπόν. Βέβαια πρέπει να γίνει πολύ άλλη δουλειά, πολύ ακόμη δουλειά θα παρακολουθήσουμε τις, ε, την κατάσταση για τον προϋπολογισμό 2012-2013. Αν έχουμε τον προϋπολογισμό όπως προτείνεται, 815 σε αρχές του χρόνου, 850 ε, σε αποθεματικό από ό,τι φαίνεται για έκτακτες ανάγκες. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, θα σας πω ότι μπορεί πολύ νωρίς, πολύ νωρίς να χρειαστεί στην αρχή του χρόνου να ζητήσουμε το αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες, γιατί βλέπουμε μια κατάσταση αποσύνθεσης στη Συρία. Χρειάζεται να προβλέψουμε τρόφιμα για τροφαρμακευτικό υλικό, να κινητοποιήσουμε δυναμικό ε, προστασίας, υποδοχής παιδιών. Ήδη, ήδη είμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας και έτσι το 2013 φοβούμε ότι Και έτσι περνάω στην παρατήρηση του κύριου Κόρτε Λάστρα. Φοβούμε ότι ε, με μείωση του προπολογισμού που προτείνουν τα κράτη-μέλη και τι συνέπειε που θα έχει αυτό, γιατί ξέρετε ότι μέχρι τώρα δεν το είχαμε το φαινόμενο, μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη λίγο πολύ διατηρούσαν ε, στο επίπεδο που είχαν τους τον προπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα όμως έχουν περικοπές, 70% περικοπεί ο εθνικός προϋπολογισμός του Βελγίου ανθρωπιστικό. Ε, το ίδιο βλέπουμε και στην Ισπανία, το ίδιο βλέπουμε και στις κάτω, στις χώρες που πάντα θεωρούσαμε πως πρόκειται για μια χώρα που αναλαμβάνει τις ευθύνες της έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Ναι, όντω το πράττουν, αλλά μας λένε ότι να δεν φτάνει. Τώρα έχουν ένα πολύ καλό υπουργό, αλλά αυτό δεν αρκεί, δεν καλύπτει την ανάγκη σε πόρους. Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν να αντιμετωπίζουμε. Και έτσι τα κράτη-μέλη όταν δεν έχουν ε, λεφτά αρκετά, τι κάνουν, στρέφονται στην Επιτροπή και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Κρυσταλίνα, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω μπορείς να κάνεις». Μα τα ίδια κράτη-μέλη όμως προσπαθούν να περικόψουν ακόμη περισσότερο τον προπολογισμό της Επιτροπής. Αυτό λοιπόν, ε, αυτή η διπλή μείωση των εθνικών και του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα έχει σημαντικά ε, σημαντικές συνέπειες, πολύ αρνητικές. Η δική μου χώρα είναι από τους μικρούς παίκτες ε, στην υπόθεση αυτή, αλλά πάντως έχει αυξήσει η Βουλγαρία τον προπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και από την άλλη μας ε, επισημαίνεται διαρκώς ότι όλες αυτές οι περικοπές και η απουσία μας από τη διεθνή σκηνή θα πλήξει σοβαρότατα την διεθνή μας εικόνα. Το ίδιο θα σας επισημάνω ότι Εάν διατίθενται χρήματα χωρίς συντονισμό, χωρίς πρόβλεψη, μπορεί τελικά αυτά τα κονδύλια που θα διατεθούν ασυντόνιστα και τα να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν ρυθμό, πρέπει να αναπτύξουμε δράση και αυτό το επισημαίνω με την ε, παρατήρηση ότι ενδέχεται να έχουμε πολύ δυσμενείς εξελίξεις και ως προς την ασφάλεια της Ευρώπης, εάν δεν αναλάβουμε δράση εγκαίρως. Για δε τα... Ε, για δε τις ε, βάσεις, θα ήθελα να πω ότι η βάση των ε, αποκεντρωμένων. Δηλαδή, έχουμε βεβαίω την προσπάθεια για την ε, καταπολέμηση του υποσυτισμού, αλλά και την προαγωγή τη αντοχή των κοινωνιών, ώστε να περιορίσουμε τα προβλήματα για το μέλλον. Πολύ καλή σχέση λοιπόν έχουμε εκεί. Κρίσιμη σημασία για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η FAO είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, ε, βέβαια το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών μεγαλύτερος, αλλά και η FAO έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα πλημμυρών, επραδείγματι, που υπονομεύουν την ευημερία των πολιτών. Άρα δουλεύουμε όλο και πιο στενά μαζί τους. Ε, πάντως θα ήθελα να πω για όποιον επένεσε το έργο μας ότι τα, οι έπαιρνοι πρέπει να πάνε στην ΕΚΟ, η Γενικός Διευθυντής είναι εδώ, αλλά πάνω απ' όλα στο προσωπικό που έχουν αναπτυγμένο στις διάφορες χώρες επιτόπου, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες που δουλεύουν ώρες ατελείωτες όταν υπάρχουν περίοδοι κρίσης και που διακινδυνεύουν ακόμα και τη σωματική του ασφάλεια και τη ζωή του όταν πάνε στι περιοχέ αυτέ. Θα το πούμε οπωσδήποτε αυτό βεβαίω. Το μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά σα. Κύριε Νιούτον Το θέμα της Σαχάρας. Ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, το λησμόνισα. Επειδή άλλαξα τη σειρά των ερωτήσεων, το χάσα. Λοιπόν, ναι, είναι μια προφανής περίπτωση κατά την οποία η περικοπή στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών έχει δυσμενέστατες συνέπειε. Εμείς διατηρούμε στο επίπεδο των προηγουμένων ετών τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια από τι λησμονισμένε κρίσεις. Είμαστε από του λίγους χορηγού που παραμένουν πιστοί και προβλέψιμοι. Ε, Βεβαίω θα θέλαμε να κάνουμε πιο πολλά, να αντισταθμίσουμε την έλλειψη από τις χορηγίες των κρατών μελών, αλλά τα περιθώρια είναι πολύ, πολύ περιορισμένα. Δεν μπορώ να σας πω πόσοι, πόσα μέλη της ομάδας με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Κύριε Επίτροπε, πρέπει να κάνουμε πιο πολλά εδώ». Ο άλλος μου λέει «Πιο πολλά εκεί, πιο πολλά παραπέρα». Είναι όμως πολύ δύσκολο με τόσες περικοπές στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, ό,τι μπορείτε εσείς να κάνετε ως Κοινοβούλιο για να διαφυλάξετε αυτή, αυτή την ευελιξία στον προϋπολογισμό και το αποθεματικό έκτακτη ανάγκης που είναι η πιο σημαντική υπηρεσία που εσείς μπορείτε να προσφέρετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε να βοηθήσουμε και ενώ προσπαθούμε να το βγάλουμε από τον τίτλο 4, επανεφέρεται στον τίτλο 4 μια παραλογική κατάσταση κατά την οποία η λεγγύη, η οποία εμάς αφορά τους Ευρωπαίους, Ευρωπαίοι να βοηθήσουν Ευρωπαίους, βρίσκεται έξω από τον προϋπολογισμό, η ευελιξία έξω από τον προϋπολογισμό, αλλά το αποθεματικό ε, έκτακτης ανάγκης, η αλληλεγγύη, την οποία, η οποία βοηθάει τους πιο φτωχούς, τους πιο δυστυχισμένους, βγαίνει και πάει στον τίτλο 4. Πρέπει να βγει εκτό προπολογισμού και ελπίζουμε ότι το κοινοβούλιο θα μα βοηθήσει να αποκαταστήσουμε τον προπολογισμό στα προηγούμενα επίπεδα. Επαναλαμβάνω, δεν ζητήσαμε για να ε, γίνει αυτό. Δεν θελήσαμε δηλαδή να κάνουμε τους Ευρωπαίους να υποφέρουν προκειμένου να έχουμε μισή πιο πολλά λεφτά. Ο κύριο Νιούτον Εγώ πρέπει να φύγω γιατί περιμένω έναν επισκέπτη, αλλά η βοηθός μου θα καταγράψει την απάντησή σας. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνει, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κίνα έχει αρχίσει να κινείται προς αυτή τη δραστηριότητα. Τι κάνουν οι ΙΠΑ, συνδράμουν. Γεωργίευα. Α, όχι, όχι, θα απαντήσω σε σειρά ερώτηση. Μίτσελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσίαση αυτή. Εμείς είμαστε, θα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 40 χρόνια και θα αποτανθώ στη γερουσία της Ιρλανδίας. Θα ήθελα λοιπόν, ε, σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ιρλανδική γερουσία, να μου πείτε τι μπορώ να προτάξω. Θα πρέπει να μπορούμε να, θα πρέπει να πούμε στο κοινό μας τι ακριβώς κάνουμε. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, θεωρούν ότι κατασπαταλούμε το δημόσιο χρήμα. Και θα ήθελα ένα δικό σας σημείωμα ως προς τη συγκεκριμένη μας δράση. Μας μιλήσατε για τα δημοσιονομικά. Θα πρέπει να μας πείτε ε, τι γίνεται ως προς την ενδεχόμενη κατασπατάληση ή μη χρημάτων. Ο πρόεδρος Σούλτς μας μίλησε σε σχέση με τη δραστηριότητα της Όλαφ σε αυτό το τομέα και την ε, κατασπατάληση. Ως προς την ε, ανθεκτικότητα όπως την ορίζεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε και τις καταστροφές δηλαδή να μειώσουμε, τη... να προλαμβάνουμε καταστάσεις ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια κυρίως, για να έχουμε λιγότερους θανάτους. Δηλαδή, αν προλάβουμε καταστροφές, θα χρειαζόμαστε και λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Κατά συνέπεια, πώς μπορούμε να ε, ενδυναμώσουμε αυτή την προσέγγιση μείωσης του κινδύνου. ως προς την έκθεση της Επιτροπής για το Συντονισμό και το γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει συντονισμός έχουμε στην ουσία απώλεια 6 δις ευρώ ως προς την εφαρμογή της αναπτυξιακής μας βοήθειας και της ε, ανθρωπιστικής. Μιλάμε για 30 δις σύμφωνα με τα δεδομένα της Κομισιόν. Εσείς είπατε 400 εκατομμύρια για τους πρόσφυγες της Συρίας, έτσι δεν μας είπατε. Και μας είπατε ποιο ποσοστό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που προσεγγίζει το ίμιση. Τι συντονισμός υπάρχει για την ανθρωπιστική αυτή βοηθή. Δηλαδή, στην ουσία πρέπει να προλάβετε την κατάσταση ή να την αντιμετωπίσετε άμεσα και όχι να κάνετε εξαγγελίες. Τι υποδομές υπάρχουν με τις ΜΚΙΟ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εξαιρετική σας ε, παρουσία, Γκέρενς. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κεωργίευα ο συνήθως τονίζει ποια είναι τα σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά είναι η κοινική, θα έλεγα, στάση την οποία ακολουθούν τα κράτη-μέλη που ετοιμάζονται για την ομιλία του τέλους του έτους, όπου θα ανακοινώσουν ένα νέο όμορφο κόσμο, ενώ στην ουσία θέλουν το αντίθετο. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουμε να απευθύνουμε εκκλήσεις προς τις κυβερνήσεις για να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει τίποτα. Οι κυβερνήσεις είναι αποφασισμένες να μας αφήσουν να διαμαρτυρόμεθα, να διαμαρτυρόμεθα, ώσπου να κουραστούμε και να σιωπήσουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια διαφορετική μέθοδο για να μπορέσουμε να τους μετακινήσουμε. Αναφερθήκατε στην ανθρωπιστική κατάσταση στο Μαλί. Θα μπορούσατε ίσως να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες ε, για την ταυτότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων στον βορρά της χώρας. Είναι τοπική, ε, μπορούν άνθρωποι εκτός Μαλή να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους ε, ανθρωπιστικές δραστηριότητες και σε αυτή την περίπτωση τι τύχης θα έχουν στην περίπτωση που υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση. Στρατιωτική παρέμβαση η οποία θα υποστηριχθεί πάνω κάτω και από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο. Αν υπάρξει μια τέτοια στρατιωτική παρέμβαση δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ανθρωπιστικών υπαλλήλων οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί εφόσον υπάρξει είπα, στρατιωτική παρέμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας εκεί. Κυρία Γεωργίευα, έχετε πάλι το λόγο. Επιτρέψτε μου. γιατί το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε επίπεδο ανθρωπιστικό, η πραγματική δράση θα έλεγα και στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν θετικά μηνύματα για την προστασία των προγραμμάτων USAID, Αμερικανικής Βοήθειας. Αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εκεί στα πλαίσια των ε, διαπραγματεύσεων με το Κόγκρέσο. Μέχρι τώρα το επίπεδο της αμερικανικής βοήθειας έχει διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα και σε επίπεδο ανθεκτικότητας των πολιτικών μας, ε, απλά υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση δύο εβδομάδων. Ανάμεσα λοιπόν στους παραδοσιακούς εισφορείς, αυτούς οι οποίοι δίδουν τα χρήματα, Υπάρχουν δημοσιονομικές πιέσεις ανάμεσα στους δωρητές και αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα προβλήματα θα έλεγα. Σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει να ακουγόμαστε εμείς περισσότερο για να πείσουμε. Μέχρι τώρα ήμασταν πάρα πολύ διακριτικοί θα έλεγα, ντρεπόμασταν λιγάκι να ακουστούμε, αλλά πρέπει να ακουστούμε και να ακουστούμε δυνατά σχετικά με τους λεγόμενους αναδυόμενους δωρητές. Υπάρχει αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κίνα, έχουν ένα πρόγραμμα βοήθειας που αναπτύσσεται ταχύτατα. Η Ρωσία έχει δώσει την αυμοδιότητα αυτή στο Υπουργείο Κατεπηγουσών Συνθήκων, όπως λέγεται. Και στη Βραζιλία υπάρχει μια κάποια αύξηση και στον αραβικό κόσμο, αλλά υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Στις περισσότερες αναδυόμενες αγορές οι αυξήσεις δεν είναι συγκρίσιμες με τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που έχουν δηλαδή κάνουν λιγότερα από όσα θα έπρεπε να κάνουν ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη. Εμείς είμαστε το 20% της παγκόσμιας οικονομίας και 50% της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η Κίνα και η Βραζιλία είναι το αντίθετο. Είμαστε δυόμιση φορές παραπάνω στο οικονομικό μας επίπεδο με τη βοήθεια που δίδουμε, είναι δυόμιση φορές παρακάτω. Η χώρα που κάνει μια τεράστια προσπάθεια είναι η Τουρκία. Εκεί συνδέεται η οικονομική ανάπτυξη με την ανθρωπιστική βοήθεια την οποία δίδουν. Και άλλες χώρες πιστεύουν ότι το κάνουν, αλλά όταν δει κανεί τα στοιχεία, τις στατιστικές, δεν φαίνεται αυτό. Η Κίνα θα πει ότι εμείς δίνουμε χιλιάδες δάνεια άτοκα αυτό γίνεται, αλλά για την προώθηση των κινέζικων συμφερόντων. Αυτό πάντως που είναι θετικό είναι ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν καταστεί διαθέσιμες πλέον τουλάχιστον ανταλλαγή των πληροφοριών αν όχι πλήρως συντονισμού. Βλέπουν οι χώρες αυτές πόσο γρήγορα αυξάνονται οι ανάγκες και θέλουν να προχωρήσουν προς τη συνεργασία μαζί μας. Εγώ πήγα στην Κίνα στην αρχή στις επαφές ήταν κάπως επιφυλακτική, αλλά θέλουν τελικά με επιστολές που μου έστειλαν μετά να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Δεν πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί και επιθετικοί απέναντί τους. Τώρα για τον αραβικό κόσμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το ενιαίο η Σαουδική Αραβία μπορεί να είναι πάρα πολύ γενναιόδορη αλλά απρόβλεπτη και δεν μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους. Τα Εμμυράτα είναι πολύ πιο ανοιχτά, πολύ πιο δεκτικά, πολύ πιο συνεργάσιμα. Έχουν μεταφράσει επίσης και τα βασικά μας έγγραφα για την ανθρωπιστική βοήθεια στην αραβική γλώσσα. Λοιπόν, εκεί είναι πιο διαθέσιμη. Λοιπόν, δύο πράγματα να πω. Πρώτον, ελπίζω τα Ηνωμένα Έθνη να ήταν ικανότερα. Αλλά πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά, θεωρούνται πολύ φιλοαμερικανοί κτλ. Ε, και δεύτερον, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε σε επαφή, να είμαστε ανοιχτοί, δεκτικοί, διαθέσιμοι επί τη βάση των αρχών της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας. βοήθεια εμείς θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους λαούς της Ευρώπης ε, το τι κάνουμε και να επενέσουμε τους λαούς της Ευρώπης για τη βοήθεια αυτή θα πρέπει να υπάρξει και επικοινωνία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα οποία κάνουμε. αν στις χώρες σας ας πούμε γίνεται μια εκδήλωση στην οποία πιστεύετε ότι μπορούμε να στείλουμε εμείς κάποιον για να σας πει το τι κάνουμε, ε, είμαστε στη διάθεσή σας. Τώρα για τον προϋπολογισμό, εννοείται τον προϋπολογισμό τον κοινοτικών ή των κρατών μελών. Ναι, στα πλαίσια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τα δημοσιονομικά και τις δημοσιονομικές προοπτικές. Κοιτάξτε, έχω δύο μηνύματα μέχρι τώρα για το MFF. Πρώτον, ότι υπάρχει μια κατανόηση για το πόσο πολύτιμος είναι ο προϋπολογισμός αυτός για την Ευρώπη. Και δεύτερον, όταν φτάσουμε στο ταμείο, κανένας δεν έχει μεγάλη διάθεση για να κάνει το τελευταίο βήμα. Εγώ θα κάνω προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες, Δεν ζητήσαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, δεν ήμασταν υπερβολικοί και ακριβώς επειδή δεν ζητήσαμε εκτατική αύξηση δεν θα πρέπει να υποστούμε και αντίστοιχες ε, δυσανάλογες μειώσεις. Γιατί ο προϋπολογισμός μας είναι μικρός. Το να μειωθεί ένας μικρός προϋπολογισμός είναι διαφορετικό από το να μειωθεί ένας μεγάλος προϋπολογισμός. Πολύ διαφορετικό. Θα δώσουμε λοιπόν τη μάχη αυτή τώρα για το απόθεμα αν μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε να παραμείνει, εσείς σαν κοινοβούλιο έχετε θα έλεγα πολύ μεγάλο βάρος γιατί είναι τμήμα του μέσου ευελιξίας. 70 εκατομμύρια σε αιτήσια βάση ακριβώς ε, ε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού είναι κάτι το ελάχιστο για σας, πολύ μεγάλο για μας. Αναφερθήκατε για ανεπάρκειες και αναποτελεσματικότητα. Ε, αφορούν μόνο το 1,1%. Εμείς είμαστε αποτελεσματικοί, ακριβώς επειδή θέλουμε να σώσουμε ζωές. Οι υπάλληλοι μας, οι υπεύθυνοι μας είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί. Έχουμε προϋπολογισμούς 300.000 ε, ευρώ και εμείς ελέγχουμε έστω και ένα ευρώ που δαπανάτε στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων. Γι' αυτό ακριβώς η αναποτελεσματικότητα αφορά ελάχιστα ποσά και ε, το επίπεδο συντονισμού το οποίο επιδεικνύουμε επί τόπου είναι υψηλωτά του επίπεδου. Γιατί, γιατί γνωρίζουμε ένα τον άλλο, συνεργαζόμαστε σωστά, προφυλάσσουμε ο ένας τον άλλο Υπάρχουν ανεπάρκειες βέβαια και αναποτελεσματικότητες σε κρίσεις. Εδώ θα πρέπει να είμαι, θα είμαι ε, κοινική. Όταν ξεκινάει μια μεγάλη κρίση όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Όλοι έστω και οι μικροί δωρητές θέλουν να πάνε εκεί να είναι παρόντες. Και μετά όταν μαζεύονται τα χρήματα στο ταμείο ξαφνικά κάποιοι εξαφανίζονται. Λοιπόν, στο Κονγκό όταν ο κόσμος πεθαίνει δεν το βλέπει κανείς πουθενά αυτό. Δεν βλέπει κανένα ανταγωνισμό ανάμεσα στους δωρητές. Τώρα για τις υποδομές ε, στο εσωτερικό της Ευρώπης έχουμε μία ομάδα εργασίας. Θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τον σωστό συντονισμό. Έχουμε μέλλον δηλαδή. Ε, σε επίπεδο διεθνές τώρα έχουμε συνεργασία με τον ΟΗΕ που είναι συντονιστής θα έλεγα. Τα πράγματα εκεί μπορεί να πηγαίνουν καλά, μπορεί και όχι. Εμείς για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία πρέπει να συνεργαζόμαστε σωστά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Τώρα, η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη λένε ότι είμαστε σπουδαίοι, αλλά λεπτά δεν δίνουμε όταν χρειαστεί. Δυστυχώς η υποκρισία είναι μία από τις πιο βλαβερές ιδιότητες του ανθρωπίνου γένους, λέει η κυρία Γεωργίευα. Τώρα έρχομαι στην ερώτηση για το Βόρειο Μαλί. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκεί είναι τοπικοί, δεν υπάρχουν ξένοι δεν υπάρχει χώρος ούτε για Ευρωπαίους, ούτε για Αμερικανούς, ούτε για άλλους Αφρικανούς. Αλλά το τοπικό προσωπικό λειτουργεί αποτελεσματικά. Συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τις κοινότητες εκεί για πολλά χρόνια και οι κοινότητες τους δείχνουν εμπιστοσύνη. Στρατιωτική παρέμβαση, προφανώς Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εκπαιδεύσει γενικά και τους στρατιωτικούς για την προστασία των, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της χορήγησης κτλ. Και θα βοηθήσει το στρατιωτικό προσωπικό. Ε, τώρα το προσωπικό του στρατού του Μαλή, το πώς ακριβώς θα τα πετύχει αυτά είναι άλλο θέμα. Τα πράγματα είναι δύσκολα μπροστά μας στο Μαλή Φοβάμαι ότι η απαγωγή ανθρώπων που εργάζονται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στις περιοχές αυτές είναι business πλέον και φοβάμαι ότι αυτές οι επιχειρήσεις ε, θα αυξηθούν, θα αναπτυχθούν εκτός και αν υπάρξει μια σωστά διατεταγμένη διεθνής δύναμη η οποία να είναι αποτελεσματική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να πείσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους στρατιωτικούς και τους ενόπλους των αφρικανικών χωρών να λειτουργούν σωστότερα σε τέτοιες καταστάσεις. Κοιτάξτε, κάθε φορά εγκαταλείπω ή ε, ε, ε, αγνοώ για, για τις καταστροφές τώρα. Εμείς ξοδεύουμε 30% του κοινοτικού προϋπολογισμού για επενδύσεις σε τομείς ανθεκτικότητας. Εμείς είδαμε ότι είμαστε πάνω από το 20% στον τομέα αυτό, στόχος το 30%, με δύο τρόπους, δράση και ε, ταυτόχρονα να αποδείξουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστά και να λειτουργήσει αυτή η γνωστοποίηση της δράσης μας προληπτικά. Είμαι υπερήφανη εδώ γιατί θα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά έχουμε θέσει τα θέματα αυτά ε, στο υψηλότατο επίπεδο στον κόσμο της ανάπτυξης. Έχουμε δημιουργήσει ένα φόρουμ, έχουμε συναντήσει σε την Άνοιξη και το καλοκαίρι με την Παγκόσμια Τράπεζα, συζητάμε τα θέματα αυτά ο πρόεδρος ε, της ε, Τράπεζας της Παγκόσμιας, ε, η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν συζητούν μόνο για θεωρητικά θέματα, αλλά για τις πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Και για πρώτη φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για χώρες ευαίσθητες σε φυσικούς σε φυσικές καταστροφές ε, διότι συνιστούν ένα παράγοντα ανασταλτικό για την οικονομική ανάπτυξη, διαρθρωτικά ανασταλτικό για την ανάπτυξη ορισμένων χωρών. Και θα πρέπει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα να βοηθήσουν. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια βελτίωση, μια μείζων αλλαγή και είμαστε πρωτοπόροι. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να τελειώσω. Ξέχασα να απαντήσω για την εξωτερική δράση. Λίγα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Και εγώ έχω ακόμα δύο συναδελφούς που ζητούν το λόγο. Αν θέλετε. Να είστε σύντομοι παρακαλώ. Κύριε Κάσμαρεκ. Πολύ σύντομα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση. Η χαλήσω να μην την υποβάλω ακριβώ ε, εκτεταμένα τώρα. Απλώ θα να επισημάνω ότι συμφωνώ με τα όσα είπατε και τα σημαντικά θέματα. Ότι δηλαδή χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της κριτικής ανάλυσης και της εκτίμησης των επιτευγμάτων, της αξιολόγηση των επιτευγμάτων. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τόσο έχει επιτύχει η Ευρώπη ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν σε μια ειδική εκδήλωση για την 20η επέτειο της ανθρωπιστικής δράσης της Πολωνίας. Πρέπει να σας πω ότι έχει επιτύχει πάρα πολλά και αυτή η οργάνωση. Η κυρία Χόισναου ήταν η αυτού του Εθνικού Οργανισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η οποία είναι ε, άτομο με αναπηρίες και όμως έχει επιτύχει πάρα πολλά να κάνει, έχει πάρα πολλά καταφέρει, έχει μεγάλο έργο να επιδείξει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι πολλοί αυτοί που κάνουν πάρα πολύ καλό έργο σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Ζολή. Και ο τελευταίο είναι ο κύριο Μπουγιάχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους αυτού τους επένου ε, που σας απίφθηναν. Ε, δύο σύντομε ερωτήσει. καταρχά στο ένα αναφερθήκατε για το SCAE. για την, ειδική υπηρεσία, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, για το Μαλί όμως θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, μια και είναι πτώση πολύ εκτοπιστέντες και μια και φαίνεται ότι αυτοί που φτάνουν στο Μπαμάκο τείνουν να επανέρχονται στις ε, περιοχές τους, έστω και υπό όρους του νόμου της Σαρία. Γιατί δεν υπάρχει επαρκής υποδοχή, δυνατότητα υποδοχής γύρω από τον Παμάκο, την πρωτεύουσα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αυτή. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία ή να δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες ως προς την υποδοχή των εκτοπιστέντων. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ για να ολοκληρώσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα εγκόμια και για την ε, αναφορά στην 20η επέτειο ε, της ανθρωπιστικής οργάνωσης της Πολωνίας. Εύχομαι και εγώ ότι καλύτερο για τους εκτοπιστέντες πρόσφυγες. Η ε, εντύπωση μου ήταν ότι παραμένουν οι ανάγκες, δεν έχουν καλυπτεί, καλυφθεί επαρκώς. Είχα μια κάπως καλύτερη εντύπωση για το τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες εκτός των συνορών παρά οι εσωτερικά εκτοπιστέντες. Από την άλλη είναι πολύ δύσκολο όταν κανείς έχει φύγει από την αιστεία του, είναι πολύ δύσκολο και να τον ε, ανέβρουμε και να δούμε τις ανάγκες του και να του προσφέρουμε βοήθεια. Πρέπει να κάνουμε πιο πολύ προσπάθεια ανθρωπιστική εκεί. Πιο εστιασμένα. Βέβαια δίνουμε και πιο, πιο πολλά χρήματα. 39 εκατομμύρια είναι η ενίσχυση για το Μαλί. Έχουμε το δικαίωμα ή μη τι άλλο να πετήσουμε αναφορέ για το πώ θα δαπανούν οι υπηρεσίε εξωτερική δράση. Ειδικά για το μαλλί με ρωτήσατε ή εν γέννη. Μάλιστα, ναι. Ήταν ε, μια ερώτηση που έθεσα νωρίτερα. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, μας προσφέρει πολύ καλή συνεργασία στις χώρες εκεί, ένα πρόβλημα. Και γιατί, γιατί εμείς έχουμε τις δραστηριότητες μας σε πολύ δύσκολες περιοχές. Και έτσι έχουμε την αντιπροσωπεία, έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, το δικό μας το προσωπικό, με κοινού στόχους. Μικρές κοινότητε εμπιστεύονται ο Μέντον, δουλεύουν πολύ καλά, έχουμε κοινούς, ε, κοινές εγκαταστάσεις μερικές φορές, αλλά χωρίς τη βέβαια δουλειά με την εξωτερική, με την υπηρεσία εξωτερική δράση ε, και οι πρέσβει επίση μα δείχνουν ε, πολύ καλό πνεύμα συνεργασία. Οι τριβέ είναι εδώ στι Βρυξέλλε, όποιε είναι. Και ε, απορρέουν από το γεγονό ότι κάποια στοιχεία αβεβαιότητας παραμένουν. Δηλαδή για κάποιους δεν είναι σαφής η κατανομή των αρμοδιοτήτων, οι εντολές, ποιος κάνει τι. Το δουλεύουμε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ψέματα και να σας πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε μια ομάδα, παραδείγματι, για την αντιμετώπιση κρίσεων, η ανταπόκριση σε που έχει θεσπιστεί και που πρέπει να πω μερικές φορές ξεπερνάει τα όρια της εντολής της με ανθρωπιστικές δράσεις. Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πάντα κακές ε, οι προθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρετε ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι οθρωμένος με καλές προθέσεις. Και πρέπει να εξηγούμε γιατί υπάρχει αυτή η διακρίση εντολών. Γιατί ακριβώς πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε μόνο ανθρωπιστική δράση, γιατί αν θεωρηθεί ότι έχουμε πολιτική τοποθέτηση, δεν φτάνουμε να αγγίξουμε τον κάθε έναν που έχει ανάγκη. Δεν μας βοηθάνε δηλαδή αν μπουν στα δικά μας χωράφια, γιατί έχει πολιτικό χαρακτήρα η επέμβαση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και αυτή η πολύ απλή μου πρόταση είναι η εξή. Τόσα πολλά έχουμε να κάνουμε. Τόση πολλή δουλειά έχει να γίνει. Ας αφήσει ο καθένας τον άλλο να κάνει τη δική του δουλειά. Εγώ να κάνω την ανθρωπιστική μου δράση, ας κάνει υπηρεσία εξωτερική δράση τη δική της δουλειά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να λύσουμε. Έχουμε ένα περιθώριο βελτίωσης ως προς την διάκριση των αρμοδιοτήτων μας, πώς βλέπει ο καθένας τη δουλειά του εδώ στις Βρυξέλλες ιδιαίτερως, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε η κάθε άστον με έχει καταλάβει, πολλές φορές έχει δηλώσει ρητά ότι αντιλαμβάνεται ποια είναι η σημασία της ανεξαρτησίας πετερότητας ε, και της αμεροληψίας ανθρωπιστικής ε, εργασίας. Αλλά μερικές φορές όταν έρχεται η ώρα κάποιοι ξεπερνούν τα εσκεμένα. Με καλές προθέσεις ίσως για να βοηθήσουν κάποιον, αλλά όταν βοηθάνε κάποιον κάνουν κακό σε πολλούς άλλους. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Για να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ε, σας δώσω κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις, Ναι, και πλησιάζουν τα, Χριστούγεννα, στο Λίβανο. Ο νεαρός Αλή μου δώσε αυτή τη ζωγραφιά. Ζωγραφιά ενός παιδιού πολύ μικρού στην ηλικία και μου εξήγησε στη συνέχεια τι είναι αυτή η ζωγραφιά. Ένα όπλο που πυροβολεί και το νεκρό σώμα του ανιψιού του, του Αμπτουλά. Μια και πλησιάζουν λοιπόν οι γιορτές, ας μιλισμονούμε τι τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν ορισμένοι άνθρωποι σε ορισμένε περιοχέ του κόσμου. Και ας ανοίξουμε τι καρδιές μας για αυτούς. Ευχαριστούμε κυρία Γεωργίαβα για τη δέσμευσή σας και εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια και να υποστηρίξουμε τους πιο αδύναμους. Σας εύχομαι καλές ε, γιορτές και ξεκούραση την οποία αξίζετε και χρειάζεστε. Nadim Mitterrand, n'est-ce pas Nous allons maintenant aborder notre 14e point à l'ordre. Λοιπόν, περνάμε στο, σημείο, στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη ε, στρατηγική στο, στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, λέει η πρόεδρος και διακόπτη.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 Σας παρακαλώ πολύ να απομακρυνθείτε όσοι το επιθυμούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ίδια διάταξη. Ο κύριος Γκέρενς είναι ο εισηγητής μας για την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών μέσα στα πλαίσια της θητείας αυτής και θα του δώσω το λόγο για να μου μας μιλήσει για αυτό τον οδικό χάρτη. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μένα είναι επανάληψη αυτό το θέμα, διότι το συζήτησα, το συζητήσαμε με τους συντονιστές. Ο δικός χάρτης λοιπόν Είμαι διορίστηκα μόνιμος εισηγητής για την συνοχή των πολιτικών μας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε δραστήριοι και να έχουμε ενεργό συμμετοχή στο τι συμβαίνει σε θεσμικό επίπεδο ως προς τη τα γεγονότα του θεσμικού επέδου και σε σχέση με αυτή την έκθεση θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια αντίστοιχη έκθεση της Κομισιόν για την συνοχή των πολιτικών μας και πρόκειται για μια συγκεφαλαίωση και μια αντίδραση ως προς αυτή την έκθεση για το τέλος της θητείας. Διότι η Επιτροπή συνήθως υποβάλλει την έκθεσή της, θα πρέπει να υποβάλλει τη συγκεκριμένη μετά το Μάιο του 2014. Δεν έχει νόημα να υπάρχει επικάλυψη, το συζητήσαμε, για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να υποβάλουμε την εργασία μας ε, προγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που θα έχουμε μέχρι τότε από τα θεσμικά, με βάση την ε, εργασία των θεσμικών οργάνων. Στη θετία αυτή θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συνοχή των πολιτικών μας. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ή οδικό χάρτη. Θα δούμε λοιπόν πώς προχωρούν τα πράγματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανατρίμηνο κατά προτίμηση εδώ στην Επιτροπή μας τονίζοντας ιδιαίτερα εάν συμφωνούμε αυτή την στενή συνεργασία με τις άλλες ε, επιτροπές, κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο γιατί ξέρουμε πόσο είναι επιφυλακτικές οι άλλες επιτροπές για συνεργασία σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα σας πρότεινα να ακολουθήσουμε την ε, καταντιμολία διαδικασία. Δηλαδή, εάν προβάλλει μια εργασία, μια δική μας, μια επιτροπή του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αντίδρασης. Έτσι θα πρέπει να κινηθούμε. Θα έρθω σε επαφή με τις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές για να τονίσω ότι θα πρέπει να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων ως προς την συνοχή με συγχωρείτε των πολιτικών μας. Να το δούμε και διαδικαστικά και από πλευράς αποτελεσμάτων καθαρά. Και όλες οι συνιστώσεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα το πρωί υπέβαλα ορισμένα ερωτήματα, ζητήματα. Να δούμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα. Πώς ε, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και συνεπείς στο διάβημα αυτό, στα άλλα διεθνή φόρα, ε, Παγκόσμια Τράπεζα, Ηνωμένα Έθνη και ούτω καθεξής. Να δούμε ποιες είναι και οι σχέσεις μας, πώς ορίζονται οι σχέσεις μας με τον Όσα που είναι πρωτοπόρος σε πολλά επιμέρους θέματα, διότι ο ΩΣΑ όρισε τις αρχικές προδιαγραφές αποτελεσματικότητας για την ανθρωπιστική βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια, με συγχωρείτε, και επειδή το θέμα έχει ξεκινήσει στον νόσα, θα ήταν σκόπιμο να δούμε και εμείς τι συμβαίνει και να δούμε πώς ορίζουν το θέμα οι εταίροι μας, Ευρωπαίοι και μη, για να έχουμε κοινά κριτήρια για το συντονισμό των πολιτικών μας. Δεν θα ήθελα να σταθώ στις λεπτομέρειες, θα τις έχετε γραπτός Σκεγράφησα την κατάσταση σήμερα το πρωί στους συντονιστές. Προτείνω λοιπόν συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συνεδριάσεις και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν συντρέχει λόγος θα ε, ορίζεται και μία έρευνα για να δούμε πώς αντιδρούν και άλλοι διεθνείς φορείς ε, για την έκθεση του ΩΣΑ σας μίλησα. Για την έκθεση που θα πρέπει να συνταχθεί μέχρι το τέλος της θητείας επίσης σας μίλησα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια, να βρούμε έναν τρόπο συνύπαρξης ε, και με τους άλλους εισηγητές για την πολιτική συνοχή, με τον άλλο εισηγητή για την πολιτική συνοχή. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ορίζονται και οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να μην έχουμε μονόλογο, να έχουμε μια αμφίδρομη σχέση και θα ορίσουμε επιμέρους θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επιτύχει αυτή η εργασία, αυτή η μακρόπνοη εργασία. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Η, κυρία Άπστρομ, η προηγούμενη συγγήτρια, ε, ήταν η προηγούμενη, η προκάτοχός μου και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, διερκής διάλογος. Θα πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί, αλλά και να έχουμε κριτικό πνεύμα ε, καθαρά ως προς τα δρόμενα για να μην επισκιάσουμε και θέσουμε σε κίνδυνο τα, τις προηγούμενες δραστηριότητες. Τέλος, θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές είναι επιφυλακτικά στη χρηματοδότηση αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και σε περίοδο ισχνών και σε περίοδο παχαίων αγελάδων. Γιατί η αναπτυξιακή βοήθεια αποτελεί μια μόνιμη συνιστόσα αποτελεί μία μόνιμη αρχή και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας πέρα από την δική μας Επιτροπή. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να επιτύχει σε αυτή την εργασία και να αναγνωριστεί η αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής και όχι μόνο ε, διαμέσου αυτής της εργασίας. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς. Και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί ο κύριος Νόμπερτ Πόπστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ συγχαίροντας στον κύριο Γκέρενς για την ε, ανάληψη της θέσης του μόνιμου συντονιστή για την ε, συνεπή ανάπτυξη. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ στενή συνεργασία μαζί του, όπως είχαμε και στο παρελθόν με την κυρία Σμίτα Μπιάστρα Ο προθεσμός ενός μόνιμου εισηγητή για μας αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, ε, συνοχή της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη. Και όπως όλοι, όλοι γνωρίζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Σας ε, διαβεβαιώνω ότι η ομάδα PSD της Γενικής μας Διεύθυνσης έχει ε, ενισχυθεί με έναν ακόμη, με ένα ακόμη μέλος. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει την εσωτερική προετοιμασία για την έκθεση για το 2013 που αναμένεται να δημοσιευθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 με τη μορφή ενός ε, εγγράφου εργασίας από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα σχεδιάγραμμα, ένα σχέδιο που θα συνοδεύεται από μια ανακοίνωση για το ρόλο των επιχειρήσεων στην προαγωγή της ε, γενικής και ανοιχτής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου θα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και έναν τομέα ε, ιδιαίτερης προσοχής και, την, ε, και τις προτάσεις μας στην ανακοίνωση. Έτσι λοιπόν, Ήθελα για άλλη μια φορά να επισημάνω ότι η Επιτροπή προσβλέπει σε πολύ στενή συνεργασία με τον κύριο Γκέρενς για τους προσεχείς, μήνες. Η ομάδα μας, η Μαρία Σταγκρίνη που βρίσκεται εδώ, Στάνκα, Στένκα, Τσουβάσοβα που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ και υποφαινόμενο, είμαστε στη διάθεσή σα να συναντηθούμε και να προχωρήσουμε σε στενή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Κύριε Γκέρενς, κύριε Κάτσιμαρακ, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για την Επιτροπή μας. Όμως, το πιο δύσκολο από τα καθήκοντα του κύριου Γκέρενς θα είναι να εξασφαλίσει τη συνέπεια την απόδειξη της σημασίας αυτών των προσπαθειών στις άλλες επιτροπές. Θα χρειαστεί και τη βοήθειά μας. Πολύ σωστά επισήμανε την επέκταση της εντολής του μόνιμου μου εισηγητή. Αλλά νομίζω ότι το κύριο ζήτημα δεν είναι τόσο η προετοιμασία στη δική μας επιτροπή, γιατί ήδη είμαστε εμείς έτοιμοι. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας σε σχέση με συναδέλφους από άλλες επιτροπές για να τους πείσουμε για την ορθή ερμηνεία της διατύπωσης συνθήκης Λισαβόνας και να τους εξηγήσουμε ότι η καλύτερη συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών αποβαίνει όφελος, είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των δικών μας πολιτικών, αλλά προς το συμφέρον ολόκληρης της Ένωσης, της αξιοπιστίας, της συνοχής και της εξωτερικής της εικόνας, της εικόνας της προς Πρέπει λοιπόν οι πάτες να υποστηρίξουμε τον κύριο Γκέρανς. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέρανς, εσείς. Ναι, Πρόεδρε. Κύριος Κάτσμαρεκ, νομίζω. Επέμεινα σε ένα σημείο πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πόσο περιορισμένη ήταν η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες επιτροπές, δυστυχώς. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και ίσως θα ήταν η λύση, η καλύτερη ενημέρωση, η παιδαγωγική δράση δηλαδή. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να επιτύχει, το είπα και νωρίτερα, παρά μόνο αν γίνεται έτσι κατά αντιμολία, έτσι ώστε ο κατηγορούμενος να είναι σε θέση, όποιος κατηγορείται για κάτι, να μπορεί να προβάλλει τα επιχειρήματά του. Αλλά ήδη, πριν ξεκινήσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διερευνούμε κάποιους Ενδεχομένου κοινού δρόμους δράση. Άτυπα. Εγώ ίσως πρώτο πρώτα αλλά και οι συνάδελφοι από τι άλλε ομάδες να έρχονται σε επαφή, καθένα με τη σειρά του, με τον αρμόδιο κάθε επιτροπής. Την πιο προφανή προσωπικότητα θα έλεγα. Φερρυπίν στην Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου. Φερρυπίν στην Επιτροπή της Γεωργία. Θα έπρεπε να του εξηγούμε ότι δεν έχουμε στόχο να θέσουμε κανένα στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αλλά να κοιτάξουμε μόνο εάν μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ή εάν κάποιες δράσεις ενδεχομένω αποβαίνουν αντιπαραγωγικές. Και έτσι αν μπορούμε να θέσουμε σε μια νέα προοπτική το επιδεκόμενο αποτέλεσμα, τότε μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι να, τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται αποδεκτά. Φερρυπίν, κοινή γεωργική πολιτική. Και εδώ ε, έμαθα για τι επιστροφέ τη εξαγωγή γεωργικών προϊόντων. Ήδη υπάρχει πρόοδο αυτό λένε οι συνάδελφοι. Το ίδιο ακούω και από την Επιτροπή γεωργία. Αλλά όταν κάθονται και οι δύο επιτροπέ να συνομιλήσουν, δεν μπορούμε να βρούμε κοινό πεδίο συνεννόηση. Ε, αυτό είναι παράλογο. Εκεί είναι που υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να προβούμε σε μια προσπάθεια ανάλυσης και βελτίωσης της συνοχής των πολιτικών υπάρχει αυτή η ανάγκη για πιο πολύ κατα... εκπαίδευση θα έλεγα, παιδαγωγική δουλειά δηλαδή προς τους συναδέλφους. Ιδιαιτέρως, εγώ ε, και ως εισηγητής βεβαίως θα ε, ενημερώσω τα μέλη των άλλων επιτροπών για τη διάθεσή σας για συνεργασία. Στον χρόνο που μας μένει, στην τρέχουσα θετία, νομίζω πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και στα όσα δηλώνουμε για να μην έχουμε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Έχετε, από ό,τι κατάλαβα, μια έκθεση το 2013. 2013, εγώ περίμενα το 2014, αλλά Το 2013 μαζί με ανακοίνωση και αυτό λίγο πολύ ανατρέπει τον δικό μου, το, δικό μου χάρτη. Άρα η δική μου έκθεση θα ακολουθήσει τη δική σας έκθεση, έκθεση Επιτροπής 2013. Αν κατάλαβα καλά ή μήπως κάτι δεν καταλάβαμε. Εγώ είπα νωρίτερα ότι περιμένω την έκθεση της Επιτροπής μετά το τέλος της τρέχουσας θητείας. Ενώ εσείς μου λέτε ότι θα καταθέσετε έκθεση 2013. Μαζί με ανακοίνωση. Άρα ο δικός χάρτης θα μπορούσε να έχει μια θεμητή βάση εν προκειμένου τα έγγραφα της Επιτροπής, έτσι ώστε να διατυπώσουμε στην Επιτροπή μας συγκεκριμένε προτάσεις. Άρα μπορούμε να πούμε ότι την κάνουμε για το δεύτερο ήμιση του 2013 και το 2014 αρχές, κάποιες, ε, σε κάποια συνεδρίασή μας, να μπορούμε να το συστήσουμε. Καλώς λέει η Πρόεδρος, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Τάιλορ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζήτω συγγνώμη. Δεν είχα καταλάβει, δεν με ενημερώθηκα ότι άλλαξε η σειρά των παρεμβάσεων και ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τον κύριο Γκέρενς. που έχω υποβάλει και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από ό,τι βλέπω πάντως, έχει προχωρήσει μεταξύ συζήτηση και μια από τις κύριες προκλήσεις είναι η απουσία συνοχής μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων της Ένωσης και των Επιτροπών. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο για να ε, βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος αυτού. Φερρυπίν ε, με μία μελέτη αξιολόγηση των συνεπειών της συνοχής της πολιτικής της απουσίας αυτής. Ζητώ και πάλι συγγνώμη γιατί ήμουν σε μια ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή Μεταφορών, έφτασα με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να τα συστήσουμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πια έχουμε, έχει κλείσει το θέμα αυτό. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Γκέρενς. Δεν θα ήθελα να απαντήσω άμεσα σε αυτό το ερώτημα σκόπιμα ετέθη. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ θεσμικών οργάνων. Για παράδειγμα, οι συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Γνωρίζουμε ότι το, το τμήμα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Κομισιόν ασχολείται με αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια συνεργασίας. Θα πρέπει να το ε, διατρανώσουμε αυτό. Δεν είναι και το μοναδικό παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο να αναλύω την κατάσταση επί δεκάμινο. Ε, φαίνεται πού μπορεί να επιτελεστεί η πρόοδος και θα ήθελα να τονίσουμε τις ε, μεγαλύτερες ανεπάρκειες που υπάρχουν και να εργαστούμε από αυτό. Ωραία. Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη τώρα. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας απέστειλε αντιπροσωπεία στην 31 η διάσκεψη της επισητιστικής ασφάλειας στη Ρώμη. Ο Ρικάρντο Κόρτες Λάστρα ήταν επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας που, όπου συμμετείχαν και η Νιούτον Ντάν και η Κέι Τέιλορ. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κόρτες Λάστρα για να μας παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα κατά τη συμμετοχή μας σε αυτή την 39η διάσκεψη για την επιστηστική ασφάλεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Γραμματεία για την υποστήριξη και την εργασία στην αντιπροσωπεία αυτή κατά τη διάρκεια των ημερών ε, που περάσαμε στη Ρώμη. Πήγαμε λοιπόν στην Επιτροπή Ασφάλειας των Τροφίμων που ξεκίνησε το 1974 σαν διακυβερνητικό όργανο με στόχο την αλλαγή των επισητιστικών πολιτικών. Στόχος είναι να καταστεί το βασικό ε, διεθνές και διακυβερνητικό φόρουμ χωρίς αποκλεισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε εγγυήσεις ε, ε, στην, στην ε, La delegación que parte... για την ε, επισητιστική ασφάλεια. Εμείς ήμασταν εκεί σαν παρατηρητές και εξετάσαμε γενικά τις απειλές για την επισητιστική ασφάλεια σε χώρες με ε, παρατεταμένες κρίσεις. Συζητήσαμε επίσης την δυνατότητα υπογραφής ενός New Deal με τις λεγόμενες έφραστες χώρες με στόχο την αποκατάσταση της τροφιμικής ασφάλειας στον κόσμο. Η αντιπροσωπεία μας πήρε μέρος επίσης και ε, στην Υπουργική Συνάντηση υπό την Προεδρία του κυρίου Λεφόλ, του Γάλλου Υπουργού Γεωργίας, για τις τιμές των γεωργικών προϊόντων, έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστότερη μορφή συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών για να διασφαλιστεί η ε, πτητικότητα σε εισαγωγικά των τιμών των τροφίμων και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες αυτών των απότομων αυξήσεων στις, ε, και να περιοριστούν στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουν ε, λοιπόν ξεκινήσει κάποιες ε, προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και στην ίδια την Επιτροπή και στο λεγόμενο σύστημα υψηλού επίπεδου για την αμοιβαία ενημέρωση για τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Ε, πήραμε μέρος και σε πολλές, θα έλεγαν, επίσημες συναντήσεις. Τέσσερις από αυτές είναι σημαντικές. Μία από αυτές είναι με την κυρία Κόσινγκ εκτελεστική διευθύντρια του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων, μία συνάντηση με τον ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Ναβάρο, μία συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή ε, της ΦΑΟ, τον κύριο Ντασίλβα, και με εκπροσώπους επίσης μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο θέμα της αποκατάστασης της επισητιστικής ασφάλειας. Βασική στόχη αυτών των, των συναντήσεων ήταν καταρχάς να δημιουργηθεί ε, μια αντιστοιχία ανάμεσα στην προσπάθεια την οποία κάνουμε ε, και στην σύνδεση της τροφιμικής βοήθειας με την ανάπτυξη. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι κάτι το οποίο μπορεί βέβαια να δημιουργήσει κάποιες δυνατότητες έτσι ώστε ε, να υπάρξει καλύτερη αποτελεσματικότητα ε, της δράσης μας. Για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός επί τη βάση αποδεδειγμένων εμπειριών και αποτελεσμάτων μέσω παραδοσιακών ε, δωρητριών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω αναδιωμένων δωρητριών όπως η Δημοκρατία της Κίνας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες απειλές επισητιστικές που προκαλούνται πολλές φορές από πολιτικά γεγονότα όπως η Αραβική Άνοιξη, αυτά που συμβαίνουν στην Συρία και στο κέρας της Αφρικής. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι και σε, μετά από επαφές που είχαμε με τον κύριο Ναβάρο έθεσε τις προτεραιότητές τους, στις προτεραιότητές τους και τις επαφές με τα κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στόχος είναι να δημιουργηθεί το ευρύτερο δυνατό κοινοβουλευτικό μέτωπο για την καταπολέμηση της ακραίας ένδυας και της πείνας και τα τρία μέρη συμφωνούν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της κατανομής των διαθεσίμων τροφίμων, κάτι το οποίο θα πρέπει να επηρεάσει και την πολιτική των δωρητριών ε, χωρών. Θα πρέπει να υπάρξει, όπως είπα και εγώ, ε, θα έλεγα μια επισητιστική δικαιοσύνη. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή θα είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύτατο πλαίσιο δυνατότατας παρέμβησης μετά από την συνάντηση στο Ρίο ΣΥΝ 20 με επιμονή στα θέματα της αηφόρου ανάπτυξης, θέματα που άπτονται του τομέα μας σε σχέση βέβαια πάντα και με τις δημοσιονομικές προοπτικές και η ανάληψη προεδρίας από την Ιρλανδία είναι μια νέα ευκαιρία. Ο κύριος Ναβάρο αναφέρθηκε επίσης ε, να υπάρξει μια διάσκεψη ε, για την αηφόρο ανάπτυξη στην Ισπανία στις αρχές του 2013 που θα έχει ένα από τους βασικούς στόχους την επισητιστική ασφάλεια. Και γι' αυτό ε, προκαλεί, προσκαλούμε στην, θέλω να προσκαλέσουμε στην Επιτροπή μας την κυρία Γκόσιν και τον κύριο Ναβάρο ε, σαν εκπρόσωποι στη συγκεκριμένη περίπτωση του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριος Τέιλορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μαζί με τον Ρικάρντο και τον Τόνι Νιούτον Ντάν ε, ήμασταν τυχεροί που πήγαμε στη διάσκεψη αυτή στη Ρώμη. Ήταν πρώτη φορά που πήγα σε μια τέτοια διάσκεψη γιατί είμαι πρόσφατος εδώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση μαζί με άλλα βέβαια και το είπε ο Ρικάρντο είναι ότι οι βασικές στατιστικές για τους ε, επισητιστικά ελληματικούς ε, κατοίκους ε, του κόσμου έχει μειωθεί στα 800 εκατομμύρια από ένα δις που ήταν πριν μερικά χρόνια. Δυστυχώς όμως τα υποσύνολα για την Μέση Ανατολή και την Αφρική έχουν αυξηθεί κατά 73 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό δείχνει τις τεράστιες προ... προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας αν βλέπουμε τις στατιστικές αυτές. Στη διάσκεψη ακούσαμε και διάφορα για τους τρόπους με τους οποίους ε, κάποιες ε, φτωχές ε, γεωργικές βασικά οικονομίες μπορούν να βοηθηθούν. Μιλήσαμε για θέματα επενδύσεων σε μικρής κλίμακας γεωργικές δραστηριότητες που είναι τρεις φορές πιο αποτελεσματικές από άλλες μορφές παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ένδυας, γιατί τα χρήματα πηγαίνουν ακριβώς εκεί όπου οι φτωχοί των φτωχών ζουν και εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα. Η διάσκεψη συζήτησε επίσης και το ρόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια των επισητιστικών κρίσεων Υπήρξε συζήτηση επίσης και για τη χρήση της αναπτυξιακής βοήθεια έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα πλαίσια της διακυβέρνησης και των υποδομών που χρησιμοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αύξηση του ΑΕΠ είναι κάτι το οποίο δεν διασφαλίζει αυτόματα την μείωση της ε, πείνας, αλλά πολλές φορές δεν έχει νόημα να, να βασιζόμαστε σε αυτό το παράγοντα. Κάποιες από τις χώρες της Νότιας Αφρικής έχουν υψηλές αυξήσεις ΑΕΠ, από την άλλη όμως βλέπουμε να υπάρχει και αύξηση των ανθρώπων που πεινούν στις περιοχές αυτές της Αφρικής. Υπήρξε επίσης αναφορά και στη σημασία της προσπάθειας ενθάρρυνσης ανάληψης μεγαλύτερων ρόλων στην οικονομία των τοπικών περιοχών από τις γυναίκες. Οι γυναίκες παράγουν τρόφιμα και έχουν, θα έλεγα, καλύτερες επιδόσεις ε, ε, επένδυσης σε κοινωνικές δομές όπως ε, η εκπαίδευση και φυσικά η ανατροφή των παιδιών. ξέρετε ότι ο πληθυσμός μας το 2050 θα φτάσει τα 9 δις. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ε, μια κάποια, θα έλεγα, σωστή μορφή προσανατολισμού των πολιτικών μας, όχι μόνο σε σχέση με το συνολικό ποσό της βοήθειας, αλλά σε σχέση με την πραγματική αξία που αντιπροσωπεύει. Και το καλύτερο το κράτησα για τελευταίο γιατί είχαμε και εκπροσώπους του Μπαν Κιμούν, δεν ήταν ο ίδιος εκεί βέβαια, μίλησε για τον στόχο της μηδενικής φτώχειας, των, των, της μη, μηδενικής και μίλησε για τις απαιτήσει που πρέπει να ικανοποιηθούν και είπε ότι ο μοναδικός ικανοποιητικός αριθμός των πεινασμένων είναι το μηδέν. Ο Νέιβιτ Ναβάρο, στον οποίο αναφέρθηκε ο Ρικάρντο, είναι ο ειδικό εκπρόσωπος του Μπαν και θα έλθει να παρουσιάσει τον στόχο πρόκληση <clears throat> στην Επιτροπή Ανάπτυξης τον Ιανουάριο. Και εγώ θα ήθελα να ζητήσω μια γραπτή δήλωση με έγκριση του Κοινοβουλίου για την αποδοχή αυτού του στόχου. Αυτά. Νομίζω ότι ήταν μια καλή διάσκεψη και είμαι ικανοποιημένος για τη συμμετοχή μου σε αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους παρευρισκομένους στην διάσκεψη της Ρώμης. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένα ζητήματα επαναλαμβάνοντας πρώτα ότι είμαι πολύ σκεπτικός ε, σε τέτοιου είδους διασκέψεις οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν ε, ε, κάποια σκοπιμότητα. Δηλαδή, ε, ίσως πρόκειται για φλιναφήματα που δεν έχουν και λόγο ύπαρξης επί της ουσίας. Ποια ήταν η θέση των υποανάπτυξη χωρών τίθεται το ε, ερώτημα σε σχέση με την υφαρπαγή γεών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες εκφράστηκαν ως προς τις διαρθρωτικές τους ανάγκες για τη δική τους δηλαδή αγροτική πολιτική. Για να αναφέρομαι για τις υποανάπτυξη χώρες σχετικά με τις απότομες αυξήσεις τιμών. Ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Είναι κάτι το αρνητικό. Τώρα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε για τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να είναι υψηλές, μεσαίες, χαμηλές. Κάθε φορά που τίθεται το ερώτημα, απάντηση δεν δίδεται θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα επαρκές ε, θα έλεγα επίπεδο αμοιβή για να παραμείνει ο Γεωργός ε, στην περιοχή του. Το θέμα είναι το επίπεδο αυτό θα πρέπει να είναι το ίδιο για όλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τη μέθοδο την οποία ακολουθούμε για να κινητοποιήσουμε τη γεωργική παραγωγή. Και τέταρτη ερώτηση, θέτω προς την Επιτροπή τη συγκεκριμένη ερώτηση, σε αυτή τη διάσκεψη στην οποία πήρε μέρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα υπήρξαν κάποιες δυνατότητες εμπλουτισμού των εταιρικών σχέσεων με τις υποανάπτυξη χώρες για την προστασία της γεωργικής παραγωγής σε αυτές τις χώρες. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κέις έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Charles Taylor, για πρώτη φορά παρευρέθην σε αυτή την ε, διάσκεψη για την επιστημιστική ασφάλεια. Γι' αυτό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Συμμερίζομαι τα σχόλια που προανέφεραν ε, οι βουλευτές. Πραγματικά ήταν ενδιαφέρουσα εβδομάδα και σκόπιμη. Για μας η διάσκεψη αυτή είναι το, ο πιο σημαντικός ε, φορέας που προωθεί την επιστηστική ασφάλεια. Και νομίζω ότι ο Οργανισμός Επιστηστικής Ασφάλειας έχει πολλούς συμμετέχοντες την κοινωνία των πολιτών, πολλούς οργανισμούς στα κράτη-μέλη και οποιοδήποτε μπορεί να προσέλθει να μιλήσει για θέματα επιστηστικής ασφάλειας. Πρόκειται για έναν ευρύτατο φορέα λοιπόν και έτσι μπορεί να διαμορφώσει τις πολιτικές επιστηστικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε ιδιαίτερα την ε, μεταρρύθμιση αυτού του φορέα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται λίγο καλύτερα στα καθήκοντά του. Ως προς το, τις τροχιλές ε, τράπεζες σε σχέση με την επισητιστική ασφάλεια, Έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, το ίδιο και για τις κλιματικές αλλαγές. Ήταν λίγο πιο προβληματικό το θέμα, αλλά τα στρογγυλά αυτά τραπέζια δεν ενείχαν πολλές ανταλλαγές απόψεων, όπως θα περίμενε κανείς. Αλλά αυτή ήταν και η πρώτη μου εμπειρία. Ε, στην ουσία έγιναν πολλές παρουσιάσεις, δηλαδή ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία τους και γι' αυτό ε, ήταν ε, κάτι το αρνητικό. Επρόκειτο για προδιαγεγραμμένες θέσεις που αναγνώστησαν και τίποτα άλλο. Επίσης, έγινε λόγος όχι μόνο για το ΦΑΟ, αλλά και για την IFAD και για τους τρεις φορείς, θεωρώντας ότι θα πρέπει να συνεργαστούν εκεί που γίνεται και να, εργάζονται καλύτερα, να συνεργάζονται καλύτερα με την ε, Κομισιόν. Οργανώθηκε δηλαδή κάτι ξεχωριστό. Ένα άλλο θέμα σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει μεγάλη σημασία να μιλάμε με μία φωνή, κάτι το οποίο ε, δεν ισχύει πάντα. Θα αλλάξει και η δήλωσή μας, θα ευθυγραμμιστεί και η δήλωσή μας ε, περί αρμοδιοτήτων σε συνεργασία με το ΦΑΟ, για να, γιατί βασιζόμασταν στην κατάσταση που ίσχυε από το 1991 μέχρι το 1995. Η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν. Πρέπει να συμφωνηθούν όλα αυτά μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν. Το ε, εξετάζει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να έχουμε μία επικαιροποιημένη δήλωση αρμοδιοτήτων και και πρακτικά ζητήματα που θα συζητήσουμε το, την Άνοιξη. Τέλος, θα ήθελα γενικότερα να πω ότι ήδη έχουμε μία ανακοίνωση για την ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Αυτό το είδαμε και κατά τη διάρκεια του θέρους και τώρα θα ασχοληθούμε για, τα, για το πρακτικό σκέλος της εφαρμογής. Επίσης συντάσσεται και μία ανακοίνωση για ζητήματα διατροφής, γιατί πολλά τρόφιμα διατίθενται, αλλά μπορεί να μην έχουν τη σωστή θρεπτική αξία. Αυτό μας απασχόλησε και πιστεύουμε ότι το κείμενο θα εγκριθεί από την Επιτροπή έτσι ώστε να έχουμε την ανακοίνωση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές ε, Μαρτίου. Άρα επί Ιρλανδικής Προεδρίας θα προωθηθεί αυτό το ζήτημα, όπως σας προείπα. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Γκέρενς, δεν μπορώ να απαντήσω. για το ποια στοιχεία ε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Επιτροπή έτσι ώστε να τα εντάξει στην ατζέντα της θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της τρεπτικής αξίας των τροφίμων. Ε, προβάλαμε μία ε, πολιτική επισητιστικής ασφάλειας το 2010, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή, κάτι το οποίο δεν έγινε άμεσα. Κατά την Ιρλανδική Προεδρία θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο για να καλύπτουμε την επισητιστική ασφάλεια γενικότερα, αλλά και το θέμα της ανθεκτικότητας και της διατροφής. Αυτά τα δύο σκέλη θα εγκριθούν ε, εκ των υστέρων. Άρα καλύπτουμε και τις τρεις αυτές πολιτικές, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει με βάση και την ε, νέα κατάσταση. ως προς τη μεταβλητότητα των τιμών και πώς ε, μπορούμε να κινηθούμε σε ένα καλύτερο μοντέλο μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας ως προς τη μεταβλητότητα των τιμών. Αν δούμε και την έκθεση του ΦΑΟ, βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο ήταν το 2008-2009 που οδήγησε και στο μέσο επισητιστικής βοήθειας. Άρα δεν χρειάζεται και η ίδια προσέγγιση γιατί δεν υπάρχει και η ίδια σοβαρότητα. Υπάρχει βεβαίως ε, μεταβλητότητα αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα ως προς την ε, επιχειρηματικότητα Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα και μέσα στα πλαίσια της επισητιστικής ασφάλειας. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις μικρές επιχειρήσεις και ε, ε αναφερθήκατε στην εργασία του David Borrow. Εγώ ε, είχα παρευρεθεί στην ε, εκκίνηση του δικτύου αυτού επιγραμμικά και ασχοληθήκαμε όχι μόνο με θέματα διατροφής αλλά και επισητιστικής ασφάλειας. Ελπίζω να απάντησα εν μέρη στο ερώτημα του κυρίου Γκέρενς. Εάν όχι να μου το πείτε. Το λόγο έχει ο κύριος Πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, ήμουν ο τρίτος βουλευτής στην αντιπροσωπεία. Στο συγγνώμη λοιπόν που αποχώρησα γιατί πήγα να δω τον ε, ε επισκέπτη μου. Τον τακτοποίησα και γύρισα. Λοιπόν, ε, είδαμε την έκθεση του Προέδρου Ρικάρντο στη Ρώμη. Έχουμε μια εξαίρετη έκθεση ε, κατάσταση και μια και έχουμε λίγο χρόνο. Είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση με την ε, Αμερικανίδα εκείνη εκπρόσωπο για το πρόγραμμα το διατροφικό και είχε συμφωνήσει όταν ε, της το ζήτησα να έρθει στην Επιτροπή να μας μιλήσει. Πιστεύω ότι οι συντονιστές θα μπορούσαν να βρουν το χρόνο να την προσκαλέσουν του χρόνου για να μας μιλήσει και για τη συνεργασία της με την κυρία Κεωργίου. Κύριε Τέλειο, ρίχτε το λόγο. Πρόεδρε, έχω αρχίσει και μπερδεύομαι εδώ. Μερική απάντηση μόνο για τον κύριο Κέρενς και την ερώτηση για την πτυτικότητα των τιμών. Θα αναφερθώ και πάλι στο παγκόσμιο Ψηφιστικό πρόγραμμα, όπως και εκείνος, όπου ε, μας εξηγούν ότι οι μικροί παραγωγοί που προσφέρουν το 50% των ε, διατροφικών προϊόντων, των τροφίμων δηλαδή στην παγκόσμια αγορά, ταυτόχρονα εκπαιδεύουν ανήκουν στην κοινωνία ε, την αναπτυξιακή ή αποτελούν ε, αναπτυξιακό δυναμικό, μπορούν να δείξουν πιο πολύ αντοχή, αιμονή, αντίσταση στις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Το ΔΕ Παγκόσμιο Πρόγραμμα έχει αναγνωρίσει τη σημασία αυτών και προσπαθεί να αναπτύξει ε, δίκτυα διατροφικά τοπικής εμβέλειας με μονιμότητα και με προβολή της τοπικής διάστασης, δηλαδή υπογραμμίζει την ανάγκη να αγοράζουμε τα προϊόντα σε επίπεδο τοπικό, να καταναλώνονται κοντά στον τόπο της παραγωγής, να μην εξάγονται, να μην κάνουν ταξίδι. Και έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά στην πιο αποτελεσματική ανά διανομή του πλούτου με την πώληση των προϊόντων, των τροφίμων κοντά στην περιοχή που έχουν παραχθεί. Να διανέμεται καλύτερο πλούτος. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα να προσπαθήσω να κλείσω επιβεβαιώνοντας αυτά που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Τέιλορ, το έγγραφο του συνεταιριστικού κλάδου και των μικρών γεωργών είναι θα έλεγα κάτι το βασικό για τις σωστές εξελίξεις σε αυτήν την Επιτροπή επισητιστικής ασφαλείας. Το είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο η ποσότητα των γεωργικών προϊόντων, αλλά και η ποιότητα και η κατανομή τους ε, σωστά. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα και αυτή είναι και η άποψη των εμπειρογνωμόνων που ήσαν παρόντες ε, στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής προσπαθούσαν να βρουν, να κάνουν προτάσεις. Ε, όχι θέμα τόσο ποσότητας λοιπόν, αλλά θέμα επιμελητίας, θέμα σωστής κατανομής, διανομής ε, των διαθεσίμων. Κάποιες απαντήσεις εδώ τώρα προς τον κύριο Γκέρεντς. Ε, για το λεγόμενο land grabbing, την υφαρπαγή γεώνα. Έχει τεθεί το θέμα μου απάντησαν ότι προσπαθούσαν να επεξεργαστούν χάρτες των διαφόρων υπήρων γύρω από το θέμα της υφαρπαγής και ότι συνειδητοποιούν το συγκεκριμένο αυτό ε, θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο τους απασχολούσε πάρα πολύ στο παρελθόν αλλά είναι ένα φαινόμενο τοπικά πολύ σοβαρό, σε κάποιες χώρες είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ενδυμικά και το θέμα δεν είναι μόνο το στο θέμα της αγοράς γεών από χώρες, ε, αλλά πολλές φορές ε, από μεγάλους ε, ιδιοκτήτες και από μεγάλες επιχειρήσεις, γεωκτήμονες και επιχειρήσεις. Τώρα για τις απότομες αλλαγές στις γεωργικές τιμές. Υπάρχουν ορισμένα μέσα τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζεται το θέμα συνεχούς επιπλέον βελτιώσεως των μέσων αυτών, έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα η πτητικότητα σε εισαγωγικά επαναλαμβάνω των τιμών. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ στα μέλη της ε, Επιτροπής, της Αποστολής και στα μέλη γενικά της Επιτροπής μας. Ήταν μια πάρα πολύ ε, θετική ε, δυνατότητα και το ότι θα έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ, του Διεθνούς, Παγκόσμιου, του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων, και την διευθύντρια του Παγκόσμιου Προγράμματος για τα τρόφιμα θα είναι κάτι το θετικό. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δεν μένει παρά να σας ανακοινώσω την ημερομηνία διεξαγωγής της προσοχής συνεδριάσεως στις Βρυξέλλες, 9η 2013, 21 Ιανουαρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και 22 Ιανουαρίου από 9 έως 12.30 και από 15 έως 18.30. Σας εύχομαι. Πολύ καλή. Πολύ καλό τέλος του 2012 και τα ξαναλέμε το 2013.